τους πολίτες της Ένωσης για την νομική ασφάλεια και για την ειχνηλασιμότητα. Όπως γνωρίζετε το θέμα αυτό είναι κάτι που θέλω να το ήθελα να, να το χειριστούμε με μεγάλη διαφάνεια σε άμεση επαφή με τους συναδέλφους, την Κομισιόν και όλους τους ενδιαφερόμενους που είναι πολλοί συνεργαζόμαστε για την ε, δημιουργία συμβιβαστικών τροπολογιών με στόχο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία θετική και επικοδομητική και που να ανταποκρίνεται στην επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου της Ναγκόγιας. Ακόμη μια φορά λοιπόν ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία μας που ήταν ενθουσιώδης και θα ήθελα επίσης καταλήγοντας να υπενθυμίσω πάλι ακόμη μια φορά τι ακριβώς παίζεται εδώ. Εδώ θα αποφασίσουμε για το μέλλον της διατήρησης της βιοποικιλότητας και δεν πρέπει να υπονομεύσουμε το κοινό αυτό σχέδιό μας για χάρη τομεακών συμφερόντων. Ευχαριστώ. Αρχίζουμε λοιπόν οι ηγητές πρώτα. Η κυρία Γκουτιέρης Κορτίνες, παρακαλώ he Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πρώτον, η Σεντρίν Μπέλια έκανε τεράστια προσπάθεια. Πολλές φορές προσπάθησε να μας πείσει με μεγάλο πάθος για τις ιδέες της και έγινε συζήτηση ανοιχτή και ειλικρινή, πολύ σημαντική. Προσωπικά αισθάνομαι μεγάλη δυσκολία και δυσφορία με αυτό το έγγραφο. Να σας εξηγήσω γιατί. Είναι λίγο προθύστερο Δηλαδή πολλές φορές κάνουμε δηλώσεις ε, για πράγματα που δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμα ή όχι. Δηλαδή το δικαίωμα σε κάτι, σε ένα στοιχείο της βιοπικιλότητας που δεν είναι πάρα πολύ καλά ταξινομημένα. Ποια είναι η χώρα προέλευσης, ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Υπάρχει μια τεράστια ασάφεια νομική ε, και ως προς το καθεστώς και ανησυχώ πάρα πολύ γιατί προτρέχουμε και δημιουργούμε μια τεράστια αβεβαιότητα αλλά και τεράστια αδικία. Γιατί καμιά φορά χαρακτηρίζουμε παράνομα πράγματα που μπορεί να μην είναι. Το πολύ πιο περιοριστικό πλαίσιο των πρασίνων έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Ε, της νομικής ασάφειας. Θα πρέπει να προχωρούμε με πιο βραδείς ρυθμούς. Να μην είναι πρωταθλήτρια κόσμου η Ευρώπη και τελικά ε, όμως να είμαστε θεροβάμονες και να μην πατάμε στη γη. Ε, γιατί έτσι εκτιθέμεθα ως Ευρώπη. Έχουμε και αδικίες. Παράδειγμα, οι αυτόχθονες λέει, εγώ είμαι πάντα ακρεφνής υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων ε, των δικαιωμάτων των ε, αυτοχθόνων. Πώς θα τους χαρακτηρίσεις ιδιοκτήτες. Ούτε δικηγόρους έχουν, ούτε τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωμά τους στα δικαστήρια. Είναι άλλη οργάνωση ένα δικαίωμα πάνω σε ένα προϊόν θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένο γραπτός νομικά ε, και από πίσω να έχεις ένα κράτος που να σε προστατεύει. Οι αυτόχθονες λαοί δεν έχουν τέτοιες κρατικές δομές για να λειτουργούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μετά υπάρχουν κάποια πράγματα ε, και κάποιες δεσμεύσει ε, με τα οποία συμφωνούμε εν μέρη. Ας πούμε θέλουμε να δημιουργηθεί κάτι, αλλά ένα ταμείο πώς θα γίνει αυτό και ποιος θα είναι ο δικαιούχος, πού θα πάνε τα λεφτά. Ακόμα δεν έχει ε, υπάρξει επαρκής ρύθμιση. Και κάτι άλλο που με ανησυχεί, δεν ξέρω αν θα εγκριθεί, είναι ο συμβιβασμός όπου ζητούμε να οριστεί τι εστί παράνομο. Όταν δεν έχει αναπτυχθεί πολύ καλά μια νομοθεσία, δεν μπορώ να κηρύττω διάφορα πράγματα παράνομα. Αν δεν υπάρχει ο νόμος που ορίζει το τι επιτρέπεται, πώς θα ορίσω εγώ τι απαγορεύεται. Μπορεί να βρεθεί κάποια συμφωνία, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη ένα κατάλογο με περισσότερη επιστημονική βάση, να δίνουμε ε, χρήματα για την έρευνα, για να υπάρχουν πραγματικοί κατάλογοι βιοπικιλότητας με επιστημονικά στοιχεία και να προχωρούμε αργά αλλά σταθερά ε, με γερά επιχειρήματα. Αυτή είναι η θέση μας και για άλλα θέματα, πρέπει να σας πω ότι καλύτερο θα ήταν να αφήσουμε ελεύθερες τις τροπολογίες χωρίς συμβιβαστικές. Γιατί αν δεν ψηφιστεί η συμβιβαστική πρόταση, χάνονται πολλές τροπολογίες που μπορεί να είναι λογικές. Μετά από αυτά που ζήσαμε χτες, δεν θέλω σε καμία περίπτωση ε, να ε, χαθεί η δεύτερη ανάγνωση. Και η δεύτερη ανάγνωση είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα που δίνει στον κόσμο την ευκαιρία να σκέφτεται και στην κοινωνία. Δεν μπορείς να τα περνάς άρον-άρον στην πρώτη ανάγνωση. Μέχρι να πάρει η είδηση ο κόσμος ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε ένα θέμα, περνάει η πρώτη ανάγνωση και έρχεται η δεύτερη και διαμορφώνεται και η κοινή γνώμη. Δεν μπορούμε όλα να τα κλείνουμε σε πρώτη ανάγνωση και να καταργούμε τη δεύτερη. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες και από τη δική μου πολιτική ομάδα που ε, χάνονται αν περάσουν συμβιβασμοί. Γενικά αισθάνομαι άβολα με όλα αυτά. Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο Χάβελ Πόκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Διότι δεν ήταν απλό το θέμα. Και απλώς να τονίσω κάποια σημεία κι εγώ. σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και τις συμβαστικές λύσεις που έχουν υποβληθεί από την εισηγητρία. Τις περισσότερες τις στηρίζω και θέλω να το πω για την έγκριση θα μπορέσουμε να το στηρίξουμε για την επακόλουθη εφαρμογή και τους σχετικούς ορισμούς και εδώ συμφωνούμε για το σύστημα των ε, πρώιμων ελέγχων και εδώ μπορώ να συμφωνήσω. Μπορεί να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως λέει και η συγκήτρια, αλλά στο συμβαστικές προτάσεις την έννοια του Ταμείου Κοινών Οφελών μπορώ να την δεχτώ Αναλόγως βέβαια πώς θα προβλεφθεί ως μέρος του προπολογισμού ή με ανεξάρτητη χρηματοδότηση. Ή θα είναι λίγο περίπλοκη διαδικασία, πάντως είναι ανεξαρτητη χρηματοδοτηση η θα είναι καλή και μπορούμε να τη στηρίξουμε. Επίσης, στηρίζω τον ορισμό των νομικώς απαιτούμενων γενετικών πόρων, της ρητής απαγόρευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως την υπέβαλε ο συνάδελφος από την ομάδα Άλντε, αλλά δεν συμφωνώ με κάποιους ορισμούς. Ιδιαίτερα για την έρευνα και ανάπτυξη που μπορεί να δημιουργήσουν αμφισημίες παραθυράκι που θα επιτρέπει σε δοκιμές να είναι μέρος όλων αυτών και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε νομίζω. Επίσης δεν συμφωνώ με κάποιες διαγραφές της παραδοσιακής γνώσης και τις σχετικές τροπολογίες που προσπαθούν να αποδομήσουν τον κανονισμό Μεταφέροντα κάποιε αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο. Εάν θέλουμε να υπάρξει μετατόπιση στο εθνικό επίπεδο, δεν υπάρχει λόγο να προωθούμε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίση για του καταλόγους και την έννοιά του όπω τις προτείνει το Έλκα έχω κάποιε αντιρρήσει. διότι νομίζω είναι εκτό πεδίου αυτού του κανονισμού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Ναγκόγια, όχι την ε, εκπόνηση νέα νομοθεσία. Σε γενικέ γραμμέ θα προτιμούσα να παραμένουμε πιστοί στο πρωτόκολλο Ναγκόγιο στο δυνατόν περισσότερο, χωρίς να εισάγουμε πολλά καινούργια στοιχεία. Να βεβαιωθούμε ότι όσα θα προτείνουμε μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι σοβαρό το θέμα. Διότι δεν χρειαζόμαστε νέες υποχρεώσεις. Θέλουμε να δημιουργηθεί ε, να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την επιστημονική γνώση στην Ευρώπη, όχι να δυσκολίες. Ευχαριστώ. Επόμενος σκιώδης είναι από την ΚΟΗ, η κυρία Λιωτάρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και πολύ καλή ήταν η συνεργασία μας με τους σκιώδεις όλους και στην έκθεσή της έχει ε, φέρει πολλές βελτιώσεις σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι' αυτό υποστηρίζω απολύτως την έκθεση. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες επίσης που έχουν κάνει πολλοί συνάδελφοι ε, και πολλές καλές ε, τροπολογίες, αλλά συμφωνώ και εγώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε να φροντίσουμε να βρούμε συμβιβασμούς για τις τροπολογίες αυτές για να συμμαζέψουμε λίγο όλο αυτό τον όγκο των τροπολογιών. Ε, ε, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα πρέπει να πληρώνονται οι ιδιοκτήτες σε περίπτωση που ε, προσφεύγει κάπου και σε αυτό το γενετικό ε, υλικό στις πηγές. Ε, το περισσότερο έχει ήδη καταγραφεί. Τώρα τι θα γίνει με κάποιο υλικό που πρόκειται να ανακαλυφθεί. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια αποζημίωση της χώρας προέλευσης. Δεν μου αρέσει αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν μου φαίνεται δίκαιη και χαίρομαι που τη βελτιώνει η συγγήτρια η πρόσβαση έχει μεγάλη διαφορά από τη χρήση στον κανονισμό. Δεν είναι μόνο η πρόσβαση, είναι και η χρήση και η γενικότερη αξιοποίηση γενετικών πηγών βάσει πρώτερης ενημέρωσης και συνένεσης με, σύμφωνη, με τα λόγου γνώσεως, σύμφωνη γνώμη. Νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για να ακολουθήσουμε το πνεύμα τη Συμφωνία τη Ναγκόγια. Και για μένα η ασφάλεια δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Το βλέπω λίγο διαφορετικά όμω από τη συνάδελφο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Νομίζω ότι οι εταιρείε και κυρίω ε, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, βοτανική τύπη, κήπη, συγγνώμη, τα μουσεία ε, τα ρυθμίζουν καλά γιατί είναι θεσμικοί οι χρήστε αυτοί. Και θα πρότεινα ε, να ενισχυθεί η δέουσα επιμέλεια στην έκθεση, ε, αυτό που ονομάζεται due diligence ε, και θα πρέπει να υπάρχει καλή ενημέρωση για να υποφελούνται όλοι οι δικαιούχοι. Έχω μια σύντομη παρατήρηση σε σχέση με την τελευταία συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών θα πρέπει να βρούμε μια λύση για τις παραδοσιακές γνώσεις, ε, για να ε, είναι στην ίδια μοίρα με τις γενετικές πηγές αυτές ε, οι γνώσεις. Και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στη χώρα για το exit και benefit sharing, πρέπει κάπως να αποζημιώνονται και αυτές οι κοινότητες με τίμιο τρόπο και σωστό για τις παραδοσιακές αυτές γνώσεις και μπορεί να γίνει με μια υποχρέωση για πρώτερη ε, συνένεση και ε, αμοιβαία ε, συνεννόηση, κάπως έτσι. Να βρούμε ένα συμβιβασμό για να αποζημιώνονται και αυτές οι κοινότητες και να μην κάνουμε τίποτα που να βλάπτει αυτόχθονους λαούς ή ε, αυτόχθονες ε, κοινότητες. Και είναι στα πλαίσια της Ναγκόγια και στο πνεύμα της συμφωνίας αυτής του 2010. Εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι την εισηγήτρια. Ευχαριστώ καρτικά. Και τώρα ερχόμαστε στους υπολείπους ομιλητές. Κρίστα Κλάς, Φρανσουάς Κροστέτς και Σοφή Οκονή. Η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ πολύ. Ακούω τη συζήτηση και βλέπω ότι πολλοί έχουμε πολλές επιθυμίες ε, για την έκθεση αυτή. Αλλά κοιτάξτε, δεν αρχίζουμε από μηδενική βάση και δεν θα πρέπει να βάλουμε τώρα σε αυτό το τσουβάλι διάφορα πράγματα τα οποία έχουν ρυθμιστεί καλά στην Ευρώπη. Η πρόσβαση στις γενετικούς πόρους, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ευρώπη ε, δεν έχει να κάνει μόνο με τη δίκαιη κατανομή των πλέον εκτιμάτων, αλλά ε, και με ευρύτερη πρόσβαση στους γενετικούς πόρους ε, και βέβαια να διατηρείται η βιοπικιλότητα και όχι απλώς να συντηρείται, αλλά να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείται κιόλας και η χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων δεν σημαίνει ότι χάνονται αυτοί. Οι χρήστε βιολογικού υλικού οπότε δεν θα πρέπει να υφίστανται επιπλέον άχρηστο και περιττό ε, βάρος γραφειοκρατικό ε, να μεταφερθεί ε, η συμφωνία της Ναγκόγια για να υπάρχει και μια καλή προστασία έχει γίνει μεγάλη ε, έρευνα ε, για τη σταθερότητα του κλίματος, για την προστασία των φυτών, όλα αυτά δεν θα πρέπει να διακυβευθούν ούτε να είμαστε εμεί μοναχικοί ε, στην Ευρώπη, στον δρόμο με τον οποίο εφαρμόζουμε τις διεθνείς συμφωνίες. Γιατί αυτό βλάπτει τους μικρομεσαίους καλλιεργητές και αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Όλοι ε, θέλουμε να αποφύγουμε τα μονοπόλια και την ε, συγκέντρωση των σπόρων και του πολυπλασιαστικού υλικού από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείε. Θέλουμε να προστατεύουμε και τους ε, αγρότες μας που καλλιεργούν και αυτοί σπόρους για ε, χρήση. Θα πρέπει λοιπόν ο ορισμός της χρήσης και του χρήστη συγκεκριμένα στον κανονισμό να είναι σαφής, σαφέστερος. Ένας αγρότης ε, που τηρεί το δίκαιο το ευρωπαϊκό αλλά έχει μια εκμετάλλευση, έχει μια καλλιέργεια και χρησιμοποιεί τους σπόρους από την καλλιέργεια για πολλαπλασιασμό των φυτών του. Άλλο είναι να χρησιμοποιείς ένα βιολογικό υλικό για πρώτη φορά και να ε, τηρείς ε, το άρθρο 4 Δεν θα πρέπει να έχουμε καταχρήσει, Έχουμε και ένα προνόμιο ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους αγρότες αυτούς. Δεν θα πρέπει ε, όμως να επεκταθεί ε, γιατί υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία και τεράστιο κόστος. Υπάρχουν τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή και θέλω και πάλι να τις ε, υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κλάς. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με όσα είπε η Κρίστα Κλάς. Ε, εάν χρειάζεται οπωσδήποτε να προστατεύσουμε ό,τι συμπεριλαμβάνει ως πλούτο η βιοπικιλότητα ως προς τα διάφορα μόρια και τα οποία δεν γνωρίζουμε ακόμη επαρκώς, έχουμε πολλά να μάθουμε και να ερευνήσουμε σχετικά, χρειάζεται βεβαίως μια ισότιμη και δίκαιη κατανομή των ωφελών με σαφεί κανόνε για την πρόσβαση. Θα πρέπει η χρήση των γενετικών πόρων να γίνεται υπό τι βέλτιστε δυνατέ συνθήκε, με υψηλέ προποθέσει ασφαλεία και βεβαίω για να διασφαλίσουμε και την διάρκεια στον χρόνο. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη βιολογική πειρατεία η οποία απειλεί τους πόρους μας ως προς το μέλλον. Και ως προς την νομική ασφάλεια θα πρέπει να δούμε τι απόφαση θα λάβουμε ως προς το κείμενο αυτό, ώστε να μην έχει και αναδρομική ίσχυ. Πρέπει να διασφαλίσουμε για τους οικονομικούς φορείς, τις μικρομεσαίες δηλαδή επιχειρήσεις, διαδικασίες ξεκάθαρες ώστε να εξασφαλίζεται η χνηλασιμότητα και να υπάρχει και δυνατότητα παρακολούθησης της αλυσίδας χρήσης αυτών των γενετικών πόρων. Θα πρέπει λόγω χάρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συντάξει έναν πρακτικό οδηγό, ώστε τα διάφορα στάδια της διαδικασίας να είναι πολύ ξεκάθαρα. Επίσης, και θα ολοκληρώσω με αυτά τα λόγια, επίσης χρειάζεται να ορίσουμε και να διευκρινίσουμε το πεδίο εφαρμογής. Το πεδίο εφαρμογής ό,τι αφορά τα, τα βασικά προϊόντα. Διότι αυτά τα βασικά προϊόντα που είναι αντικείμενο ελεύθερης πρόσβασης δεν θα πρέπει να καλύπτονται. Και ως προς αυτό να τονίσω ότι οι τροπολογίες ε, του κυρίου Γκαστον Φρακό οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση κατά την απόψη μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Κονή. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε, διότι οι συνάδελφοι ήδη κάλυψαν πολλά από τα στοιχεία που ήθελα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μπελιέ για το έργο της και να πω ότι είναι εδώ δύο τα μείζωνα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα η απλούστευση και η σαφήνεια του κειμένου, αλλά πάνω απ' όλα η ευκολία της πρόσβασης για τους χρήστες. Ε, έχουμε σωστά ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, διότι πρόκειται για στοιχεία που συχνά ε, αποτελούν κείμενο επίκρισης. Απλουστεύουμε λοιπόν τις διαδικασίες και τις παρουσιάζουμε με σαφήνεια. Ε, το ίδιο το κείμενο δηλαδή στους παραλήπτες του. Και το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως και η Κρίστα Κλάς, ότι η διάσταση των διαδοχικών χρηστών δεν θα πρέπει να ξεγλιστράει από αυτές τις διατάξεις σε σχέση με τους τελικούς ή τους μετα... μεταγενέστερους χρήστες. Να εξηγήσω τι εννοώ. Οι διατάξεις σε γενικές γραμμές είναι εύλογες, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ερμηνεία στο γεωργικό τομέα και όλος ιδιαίτερο στον τομέα των ε, σπόρων. Θα πρέπει εδώ να φροντίσουμε να διατηρηθεί η θητική ποικιλία και η, η για την επιλογή να αξιοποιούν τους γενετικούς πόρους, με συγκεκριμένους κανόνες για την πρόσβαση και την κατανομή βάσει του κανονισμού όπως θα υιοθετηθεί. Όμως, από την άλλη, θα πρέπει οι μεταγενέστερες υποχρεώσεις για τους γενετικούς πόρους και σε κάθε μεταφορά τους να μην ξεχνάμε ότι αφορούν πόρους που δεν βρίσκονται πια στην αρχική τους κατάσταση αλλά έχουν αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως. Θα πρέπει η διάταξη αυτή στην τροπολογία 40 που υπέβαλα ε, και 39 της κυρίας Κλάς που είναι πολύ παρόμοιες να ληφθούν υπόψη διότι εδώ προτείνω στην εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές μας να το μελετήσουν το, σημείο, το, το θέμα αυτό. Είμαι στη διάθεσή τους να τους εξηγήσω πόσο είναι πραγματικά κεφαλαιόδου σημασία και αναγκαίο ή υποχρεώσεις και απαιτήσει που θα προκύψουν για τους διαδοχικούς χρήστες βάσει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια να μην ακυρώσουν ουσιαστικά την ελεύθερη κυκλοφορία των φυτικών ποικιλιών ως πηγών ποικιλότητας για την έρευνα και για την βελτίωση των φυτικών καλλιεργειών με κάποιες εξαιρέσεις. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους, ε, να επενέσω και εγώ την εισηγήτρια. Πραγματικά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και προσπαθεί να βρει ένα κοινό έδαφος να προχωρήσει η Επιτροπή μας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Ποκ, τον δικό μας σκιώδη εισηγητή, τον σοσιαλιστών και δημοκρατών, γιατί πραγματικά επέδειξε ένα πνεύμα συνεργασίας και πολύ επικοδομητικό για να βρεθεί όντως ένα κοινό έδαφος και ένα κοινό πνεύμα συνεργασίας. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνένεση που έχει δημιουργηθεί γι' αυτό το θέμα της βιοπειρατείας, ε, τη δημιουργία του απαραίτητου αυτού ταμείου και επίσης την υποχρέωση για την προηγούμενη συνένεση κατόπιν ενημέρωσης για ε, καινοτόμες και περαιτέρω χρήσης ε, υφισταμένου γενετικού υλικού. πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι ε, κάτι που απασχολεί πάρα πολύ και τους πολίτες μας, αλλά είναι και κρίσιμο για το μέλλον. Για ποιο λόγο. Διότι είμαστε τώρα σε μια φάση όπου δίνουμε όλο και περισσότερα δικαιώματα ε, στις εταιρείες να κατοχυρώνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα. Αυτό κατά κάποιο τρόπο έρχεται τώρα να εξισορροπήσει τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζονται τα δικαιώματα των επιχειρήσεων για να μην είναι υπερβολικά και καταχρηστικά. και διαφυλάσσουμε και ε, κάποιες γνώσεις πρώτερες, κάποια πράγματα που είχαν ανακαλύψει ορισμένοι πριν εφερβερθούν ε, τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να είμαστε στραμμένοι προς το μέλλον και να αποφύγουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη. Σας ευχαριστώ όλους και είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα μας κάνει όλους περήφανους. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ποιος θέλει. Παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη. Ξέχασα έναν συνάδελφο. Το Ρίχαρτ Ζέμπερ. Συγγνώμη που ζητώ τόσο αργά το λόγο. Ε, νόμιζα ότι ήμουν στο κατάλογο. Χαίρομαστε που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά θα παρακαλούσα να τηρήσουμε τη νομική βάση και το πρωτόκολλο του Ναγκόγια. Δηλαδή ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να λάβουμε και άλλα μέτρα επιπλέον της Συμφωνίας Ναγκόγια, πρώτον δεν μας βοηθάει πάρα πολύ και πάλι ερχόμαστε και ζητάμε ταμείο σε, σε όλα τα νομοθετήματα ξεφυτρώνουν ξαφνικά παντού τα μία. Και πώς θα τα διαχειριστούμε αυτά μετά και τι θα τα κάνουμε. Και πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι τα, τους πόρους και τα χρήματα που θα συλλέξουμε θα τους μοιράσουμε με δίκαιο τρόπο. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα γιατί υπάρχουν και πολυμερείς συμφωνίες, αλλά οι πολυμερείς συμφωνίες δεν είναι για μας νομική βάση. Γιατί εγώ βλέπω και νομικά και τεχνικά προβλήματα. Να μην το παρακάνουμε. Ε, είμαστε τρομερά παράτολμη μάλιστα στην Ένωση με αυτό το θέμα. Προσοχή, μην χάσουμε το στόχο μας. Μην το παρακάνουμε από τον πολυζήλο. Ευχαριστώ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σάλε, παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεται να απαντήσουμε σε ορισμένα από τα προβλήματα που τέθηκαν. Πρώτον εκτιμούμε ιδιαίτερα το χρόνο και την προσπάθεια που αφιέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του, των ευρωπαϊκών προσπαθειών για τη διατήρηση και διασφάλιση της βιοπικιλότητας με βιώσιμο τρόπο. Η βασική φιλοσοφία της πρότασης της Κομισιόν είναι να προταθούν μέτρα απαραίτητα, που είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν σε ενωσιακό επίπεδο. Στο πρωτόκολλο της Ναγκόγιας υπάρχουν τρεις τομείς. Ένας η νομοθεσία για την πρόσβαση. Για μας ήταν σαφές ότι το θέμα αυτό αφορά τα κράτη-μέλη και τις δικαιοδοσίες τους. Άλλος τομέας η ισόνομη συμμετοχή στα ωφέλη όλων αυτών και αυτό είναι θέμα συμβατικών υποχρεώσεων και άρα το αφήνουμε και αυτό και το τρίτο μέτρα για τους χρήστες. Αυτό βασιστήκαμε. Χαιρόμαστε που οι περισσότεροι βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της αυστηρής εφαρμογής των νομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρωτόκολλο της Ναγκόγιας και πιστεύω ότι γι' αυτό χρειάζεται να, δούμε, να σκεφτούμε πολύ καλά τι ξεπερνάει το πρωτόκολλο αλλά επίσης και τι κινδυνεύουμε να μην εφαρμόσουμε πλήρως από αυτά που προβλέπει το πρωτόκολλο. Άρα ως Κομισιόν μας ανησυχούν διάφορα αιτήματα που ακούστηκαν για εξαιρέσει συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών ή από το πεδίο εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Είναι φανερό ότι με την εξαίρεση συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών. Τελικά αυξάνουμε την νομική αβεβαιότητα και ασάφεια. Γιατί θα πρέπει κάθε φορά να ορίζουμε αν η χρήση που κάνουν είναι εντός ή εκτός των προβλεπομένων από το πρωτόκολλο. Και αυτό οποιοδήποτε χρήστης ούτως ή άλλως πρέπει να το διτάξει μόνος του. Εμείς του το διασφαλίζουμε. Αν καταλήξουν τελικά ότι οι πόροι που χρησιμοποιούν βγαίνουν από το πεδίο εφαρμογή του πρωτοκόλλου τότε θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που παράγουν θα τηρούν τις προδιαγραφές. Επίσης οι χρονικοί, μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα γιατί μιλούμε για γενετικούς πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί από Ευρωπαίους χρήστες νόμιμα χωρίς όρους, ιδιαίτερους όρους ή μπορεί να πρόκειται για τη δημιουργία υποχρεώσεων που περιορίζουν τη δυνατότητα χρήσης αυτών των πόρων. Αυτό δεν θα ήταν καλό. Και θα αντετίθετο και στη σόφρονα θέση που πήρε προηγουμένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ένωση όταν δεχόταν την εφαρμογή της συμφωνίας. Επίσης δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι χρειάζεται απαγόρευση. Και άρα δεν βλέπουμε και κανένα λόγο να καθοριστεί, να οριστεί ο νόμιμος ή μη χαρακτήρας ορισμένων χρήσεων γιατί οι χρήστες στην κανονική δουλειά τους πρέπει εκείνοι να γνωρίζουν αν οι πόροι που χρησιμοποιούν οι είναι μέσα στο πεδίο εφαρμογής του πρωτοκόλου ή όχι. Για μας θεωρούμε ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την ερμηνεία ρητρών που αφορούν το άρθρο 4 και 5 του πρωτοκόλου της Ναγκόγιας και γι' αυτό όπως είπα και πριν οι πιθανές δυνατές εξαιρέσεις πρέπει να παραμείνουν στο ελάχιστο. παρά το ότι δεν το είπαν ρητά οι βουλευτές πρέπει να το πω εγώ ότι επιμένουμε ιδιαίτερα στα εργαλεία που προτείναμε, τα μέσα που προτείναμε μικρά εργαλεία για να διευκολύνουν τα διοικητικά άχθη των χριστών μέσω της αναγνώρισης βελτίστων πρακτικών και των λεγόμενων Trusted Collections. Γιατί χρήστες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν αυτά τα εργαλεία και που θα τους διευκολύνουν πολύ, θα είναι πολύ πιο φιλικά προς τον χρήστη. Αυτά λοιπόν τα δύο εργαλεία θα διευκόλυναν πολλούς χρήστες να εφαρμόσουν τις ρήτρε του κανονισμού πιο αποτελεσματικά και πιο φτηνά. Δεν θα θέλαμε λοιπόν να διαγραφούν αυτά γιατί θεωρούμε ότι δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους χρήστες αλλά αντίθετα διευκολύνουν τον στόχο της διατήρησης και βιώσιμης χρήσης της βιοπικιλότητας και των γενετικών πόρων στην Ευρώπη. Νομίζω αν δεν απατώμε ότι θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση, διευκρινιστική από τον συνάδελφο Γκερμπράντη, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά τους και τις τροπολογίες. Τα σχόλια για τις τροπολογίες δηλαδή. Έχω μια ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπατε. Είπατε ότι ορισμένε τροπολογίε αντιτίθεται στο πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Και ρωτώ, και τι θα μπορούσε να συμβεί νομικά σε περίπτωση που εγκρίνουμε ένα κείμενο το οποίο νομικά είναι αντίθετο με το πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Τι θα γίνει. Ε, θα υπάρξει καμιά νομική δίωξη από κανέναν. Από ΜΚΟ, από το CBD, ε, ποιες θα είναι οι συνέπειες αν ψηφίσουμε κάτι τέτοιο. Um, Παρακαλώ. Το πρωτόκολλο προβλέπει ένα πλαίσιο εντός του οποίου οι επόμενοι ε, συμβάλλοντες στο πρωτόκολλο της Ναγκόγια θα μπορούν να προστατεύσουν τους ε, γενετικούς πόρους εντός της δικαιοδοσίας τους. Αυτό όμως θα παραμένει στην ελεύθερη κρίση των υπολοιπών συμβαλωμένων στον πρωτόκολλο να καθορίσουν τι προποθέσει πρόσβαση στου δικού του γενετικού πόρου. Η πρόσβαση στου γενετικού πόρου, όπω υπόθηκε και από του διαπραγματευτέ μα ε, επανειλημμένω, η πρόσβαση θα βασίζεται στο εάν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι η δικαιοδοσία του χρήστη μπορεί να εφαρμόσει πλήρως τις συνθήκες της Ναγκόγια και αν τα πολιτικά μέτρα που έχουν ε, προβλεφθεί είναι επαρκή για την υλοποίηση του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρηθεί ότι δεν έχει υλοποιήσει πλήρως τα μέτρα συμμόρφωσης των κριστών σε πρώτη φάση, αυτό βεβαίως θα ε, επηρεάσει την προθυμία των εταίρων μας να επιτρέψουν πρόσβαση στους δικούς τους πόρους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εμπορευμένους της. Στο άμεσο μέλλον δεν προβλέπω ένομα μέσα να κινηθούν εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένδικα μάλλον μέσα, στο πλαίσιο του πρωτοκόλου της Ναγκόγια, όμως στο μέλλον, εάν υπάρξει διαδικασία μη συμμόρφωσης, μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου αν θεωρεί ότι δεν, είμαστε, δεν συμμορφούμεθα με τις ε, υποχρεώσεις μας βάσει των άρθρων 14, 15, 16, 17 και ακολούθως, τότε θα μας βάλουν στάμπα διεθνώς ως ε, μιας δικαιοδοσίας που δεν ε, έχει υλοποιήσει πλήρως το πρωτόκολλο. Με όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους. Παγκοσμίω. Ευχαριστώ, για να κλείσει, παρακαλώ. Αν θέλετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συντομότατα, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους και έπειτα να τους πω ότι συμμερίζομαι την ιδέα ότι η νομική βάση είναι προφανώς το πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Ε, Βάσει αυτής της ιδέας ε, εκπώνησα και ολόκληρη την έκθεση. Ε, για όσους είπαν ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια, εγώ να πω ότι θα πρέπει να απευθύνω, να απευθύνω έκκληση να μην υποβαθμίσουμε τα όρια του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, να μην υπαναχωρήσουμε σε σχέση με όσα προβλέπει, διότι αυτό θα μας κάνει λιγότερο αξιόπιστο σε διεθνές επίπεδο και θα μειωθεί η εμπιστοσύνη των άλλων κρατών που είναι συνεπλημένα στο πρωτόκολλο. Για πρόσβαση σε πόρους που αυτό το κανονισμό δεν διευκρινίζει απαραίτητος. Να φροντίσουμε λοιπόν να μην μείνουμε μόνο στο γράμμα του πρωτοκόλλου τη Μαγκόγια και προκαλέσουμε νομική ανασφάλεια. Άλλωστε με την τελευταία παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστη σαφέ ότι και αυτό ισχύει. Επίση, κάποιοι εξέφρασαν ανησυχίε, ιδίω οι συνάδελφοι Κλά και Οκονή, και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε αυτά που μα επεσήμαναν. Εγώ επαναλαμβάνω ότι είμαι πρόθυμη να εξευρεθούν συμβαστικέ λύσει και ως προς την ε, προθεσμία και την απέτηση που δικαιολογεί ακριβώς την αναζήτηση συμβαστικών λύσεων και εδώ απαντάω στην κυρία Γκουτιέρες Κοτίνε, ότι η οποία προτιμούσε να έχουμε περισσότερο χρόνο και έγκρισε στη δεύτερη ανάγνωση να θυμίσω το δικό μας χρονοδιάγραμμα επόμενη συνεδρία των μερών ε, το φθινόπωρο του 2014 Οπότε καλό είναι να υπάρχουν ήδη κανονισμοί για να μπορούμε να φτάσουμε στο δημοκρατικό τραπέζι με κάποια χαρτιά στα χέρια μας. Και τελευταία είδηση, κάτι που δεν είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση, 18 κράτη σήμερα έχουν εγκρίνει, κυρώσει το πρωτόκολλο και η γραμματεία της σύμβασης της επικοινότητας μας είπε ότι 33 ακόμη θα το έχουν εγκρίνει στο τέλος της χρονιάς και το τον Ιούλιο το 2014 53 συνολικά. Χρειάζονται 50 για την ε, εφαρμογή του και αυτά τα κράτη δεν συμπεριλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν διακινδυνεύουμε και επισημένω στους συναδέλφους και αυτό το στοιχείο, εάν δεν κινηθούμε με ταχύτητα και δεν περάσουμε στην κύρωση και την ε, υλοποίηση του κανονισμού όπω τον πιο σύντομα, ε, διακινδυνεύουμε να μην είμαστε στις διαπραγματεύσεις παρόντες όταν θα διευκρινιστούν πια οι όροι εφαρμογή του πρωτοκόλου σε, διεθνές ε, κλίμακα, σε διεθνή κλίμακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Προθεσμία για τις απολογίες 24 Μαΐου, 12 το μεσημέρι έχει λήξει. Στις 4 Ιουλίου θα ψηφίσουμε εδώ. Στην Ολομέλεια δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα πάει πολλά κρύβονται πίσω από αυτόν τον περίφημο τίτλο και εκπλήσουμε που είναι τόσο μικρή προσέλευση. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι από τις άλλες επιτροπές δεν κατάλαβαν καν από αυτό το γρίφο τι κρύβει ο τίτλος. Και για κάποιους άλλους κλάδους ε, και άλλες επιτροπές μας περιμένει μεγάλο κέφι σε αυτή την έκθεση πιστεύω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο σημείο 17. Είναι του κυρίου Ρώση το θέμα, ο εισηγητής μας, και του δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία, του συναδέλφου Ριβαζή Σόμαρ και Τέιλορ, οι οποίοι συμμετείχαν στις ε, φάσεις επεξεργασίας και σύνταξης του κειμένου με πραγματικά πολύτιμες ε, συνεισφορές από μένα τον ίδιο. Συνεργάστηκαν όμως και στην διοργάνωση του workshop, του εργαστηρίου που σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Σε σχέση με το θέμα αυτό να πω ότι είναι ευαίσθητο, διότι μας αφορά όλους ε, καλός ή κακός. Διότι για λόγους λιγότερο ή περισσότερο σοβαρούς, σε ένα νοσοκομείο θα πάμε. Ε, στο νοσοκομείο λοιπόν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο ασφαλή, υγιή και ότι από εκεί φεύγουμε θεραπευμένοι. Σήμερα όμως ε, και ακόμη και στα μέρη τα οποία εγώ προέρχομαι υπάρχουν κράτη από που είναι λιγότερο ή περισσότερο προσεκτικά ε, σε θέματα αυτά και βεβαίω τα πράγματα αλλάζουν και στα εσωτερικό ενό κάτω μέλου από γεωγραφική περιοχή σε γεωγραφική περιοχή και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Εδώ το κείμενο μιλάμε για 37.000 Ευρωπαίους πολίτες που κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από λοιμώξεις τις οποίες ε, έχουν ρωλήσει σε νοσοκομιακή ε, περίθαλψη και μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που έχουν ήδη τυχιακογής και έχουν θεραπευτεί. Δεν μιλάμε λοιπόν για άτομα τα οποία είχαν ιδιαίτερα προβλήματα ή βλάβες από από σοβαρέ ασθένειε. Μιλάμε για ανθρώπου που μπήκαν μια-δύο μέρε στο νοσοκομείο και 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ετησίω αφορά το θέμα αυτό. Του οποίου, όπω είπα, 37.000 ε, κατά μέσο όρο έχουν σοβαρέ ε, βλάβε οι οποίε οδηγούν στο θάνατο. Τι έχουμε κάνει και τι έχει κάνει το Συμβούλιο λοιπόν για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα για τον κανόνα και θα πρέπει να υιοθετήσουν τα κάτι μελη μας φάνηκε σχεδόν γελίο και με το είπαν και οι εμπειρογνώμονες ότι το μεγαλύτερο μέρος των λοιμόξεων ε, προκύπτουν από τον εξή λόγο. Οι γιατροί και οι νοσοκόμοι δεν πλένουν τα χέρια τους περνώντας από τον ένα ασθενή στον άλλο ή χρησιμοποιώντας εργαλεία ε, χωρίς να τα αποστηρώνουν. Αυτό φαίνεται τελείως παράλογο. Θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτή η πηγή λοιμόξεων με λίγη περισσότερη προσοχή, μηδενικό είναι το κόστος. Αρκεί το ιατρικό προσωπικό να ήταν λίγο πιο προσωπικό. Το προσωπικό των ε, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και νοσοκομείων. Με την εκπαίδευση του προσωπικού λοιπόν και την πληροφόρηση των ασθενών, διότι μιλάμε για δύο διαφορετικές κατηγορίες ως τώρα. Ο ασθενής που έχει ε, μολυνθεί από την εσφαλμένη ας πούμε συμπεριφορά του προσωπικού ή υπάρχουν παλιές υποδομές και δεν γίνεται αρκετά καλή αποστήρωση των ε, σιδερένιων εργαλείων ή άλλα ε, επιθετικότερα στοιχεία τα οποία αφορούν τα ιατρικά εργαλεία αλλά μετά υπάρχει και ο ρόλος των ασθενών οι οποίοι ο οποίος καλόπιστα υιοθετεί συμπεριφορές χωρίς να δίνει ιδιαίτερη προσοχή ε, σε κάποια στοιχεία, τα οποία μπορεί να του προκαλέσουν ε, λίμωξη. Όχι μόνο στο νοσοκομείο, αλλά και αμέσως μόλις επιστρέψει στην κατοικία του. Άρα λοιπόν, ε, εκπαίδευση του προσωπικού και πληροφόρηση του ασθενούς. Ο ασθενής έχει από τη μια το δικαίωμα να γνωρίζει ότι αν προκύψει βλάβη κατά την ανάρρωση στο νοσοκομείο, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την βλάβη αυτή και πρέπει αμέσως να αποζημιωθεί. Από την άλλη πρέπει και να γνωρίζει ότι όταν ε, είναι στο νοσοκομείο και καταλήξει ε, στην αποθεραπεία, όπου θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη, εάν δεν υπάρχει κάποιο οικογενειακό μέλος ή κάποιος που τον συνοδεύει, εκεί θα πρέπει να ακολουθηθούν ούτως ή άλλως κάποιοι κανόνες. Αλλιώς μπορεί να προκύψει πάλι βλάβη ή να ε, προκύψει λίμωξη και μπορεί να ξαναγυρίσει στο νοσοκομείο και να υποβαθμιστεί η σωματική του κατάσταση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το πούμε, γιατί δεν είναι αρκετά προσωπικά το προσωπικό των ε, νοσοκομείων ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ε, Επίση, με τι περικοπέ στα κράτη μέλη, στι περικοπέ των προπολογισμό του, υπάρχει μείωση του ιατρικού προσωπικού. Οι, οι βάρδιε του ιατρικού προσωπικού πολλέ φορέ είναι απάνθρωπε στη διάρκεια ή δεν δίνεται η επαρκής ε, προσοχή στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και άλλων ε, παρόμοιων θεμάτων. Οι προτεραιότητες λοιπόν που έχουμε θέσει είναι να αναζητήσουμε την δημιουργία να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και να προβλέψουμε ανταλλαγή των βέλτιστων δυνατών πρακτικών μεταξύ των Ιδρυμάτων των Κατών Μιλών, των κέντρων ελέγχου των λοιμόξεων και νόσων, των νοσοκομιακών λοιμόξεων κυρίω, την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών, την πληροφόρηση μάλλον των ασθενών, και επίση να μην υπάρξουν περαιτέρω περικοπέ στα κονδύλια που προβλέπονται για την υγεία. Ακόμη να επιδιώξουμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο των Νόσων και Λοιμόξεων. Μιλάμε εδώ για το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το ΕΚΠΕΝ, και για να καταμετρήσουμε τον αντίκτυπο των λοιμόξεων και νόσων τώρα, που πολλές φορές δεν έχει ληφθεί αρκετό υπόψη, αλλά θα πρέπει να διατεθεί και να ληφθεί υπόψη από τα κράτη-μέλη στο μέλλον. Δεν ίσχυουν όλα αυτά με τον ίδιο τρόπο για όλα τα κάτι μέλη, αλλά είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρο. Σα είπα, μιλάμε για 4 εκατομμύρια Ευρωπαίου που νοσηλεύονται ετησίω και ε, έχουν κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια τη ανάρρωση στο νοσοκομείο από λίμωξη. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στην έρευνα και στην ασφάλεια των ασθενών με τι βάσει δεδομένων και με τρόπο ώστε να προσφέρουμε τι καλύτερε δυνατέ υπηρεσίε στου ανθρώπου που πηγαίνουν ω το νοσοκομείο και νοσηλεύονται, που θα πρέπει να γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλέ περιβάλλον και από που δεν θα πρόκειται με μια επιπλέον ε, ασθένεια από αυτήν για την οποία πήγαν για να θεραπευτούν στο νοσοκομείο. Για του συναδέλφου ε, με του σκιώδει εισηγητέ, ήδη έχουμε προβλέψει μια σειρά από τροπολογίε, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο χαρακτήρα ε, των μέτρων αυτών δεν επιτρέπει πάρα πολλές προτάσεις, υπάρχει περιορισμός. Ε, οι συνάδελφοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν τις τροπολογίες τους ε, και θα φροντίσουμε να τις συζητήσουμε γιατί είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο δεν αφορά τις πολιτικές ε, προσχωρήσεις και παρατάξεις, αλλά είναι ένα θέμα του κοινού συμφέροντος των πολιτών μας. τώρα. Η κυρία Ζόμερ, πρώτη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή. Είναι πολύ καλή η έκθεση, το σχέδιο και το θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Να αναφερθώ σε διάφορα σημεία. Πρώτον, οι ε, λοιμώξεις που προέρχονται από τη θεραπεία, που συνδέονται με τη θεραπεία. Έχει πει πολλά και ο εισηγητής ήδη. Αυτό το θέμα θεωρώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί γιατί αυτές οι λοιμώξεις ευθύνονται ε, για όλα τα επεισόδια, κατά ένα τέταρτο των, όλων των επεισοδίων και οδηγούν σε 37.000 θανάτους το χρόνο δεν είναι αμεληταία αυτά τα μεγέθη και στη Γερμανία, τη χώρα μου, είναι πάρα πολύ κακή η κατάσταση. Αν δούμε τι γίνεται με την αντοχή των ε, μικροβίων στα αντιβιωτικά και στις κάτω είναι 1%, στη Γερμανία είναι 20% των ασθενών που εμφανίζουν ε, τέτοια αντίσταση στα βιωτικά. Ε, έχουμε ακόμα να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα ένα από τον άλλον στα κράτη-μέλη. Και βέβαια η πρόληψη θα πρέπει να είναι σε πρώτη θέση. Αλλά κάτι άλλο και σωστά το ζητεί ο εισηγητή, θα πρέπει να είμαστε και υπέρ και να φροντίσουμε για τη διαφάνεια. Δεν επιτρέπεται ο φούρναρης της γειτονιάς να διαπομπεύεται στο ε, διαδίκτυο αν μπήκαν ένα μυρμήγκι στο κέικ, ενώ τα ε, νοσοκομεία να τα κουκουλώνουν ε, όλα τα κακό σκήμενα και τα στρεβλά που συμβαίνουν. Δεν επιτρέπεται αυτό, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος για την υγεία των πολιτών και υπάρχουν χώρες που δεν τολμάει κανείς να πατήσει σε νοσοκομείο. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνεται καλύτερα όχι μόνο οι ασθενείς αλλά και το συγγενικό τους περιβάλλον. Ε, και αυτό ζητάει ο συγητής, αλλά θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με αυτό πρέπει να δούμε και τη δημογραφική εξέλιξη στην Ευρώπη. Ο κόσμος ε, γυράσκει όλο και περισσότερο και οι πιο ηλικιωμένοι ασθενείς σήμερα πρέπει να παίρνουν ταυτόχρονα πολλά φάρμακα γιατί τους τα συνταγογραφούν και τους ξεπερνάει ο αριθμός των προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνουν όταν ε, παίρνουν διάφορα φάρμακα μαζί. Ε, στη Γερμανία, για να σας δώσω έναν αριθμό, Σύμφωνα με μια μελέτη, 5% όλων των εισαγωγών στα νοσοκομεία έχουν να κάνουν με ε, ε, ατυχήματα από τη λήψη φαρμάκων. Γιατί ο κόσμος παίρνει ταυτόχρονα τόσα πολλά φάρμακα, κάνει λάθη και μετά καταλήγει στο νοσοκομείο. Ε, και θα πρέπει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των φαρμάκων που μπορεί κανείς να παίρνει ταυτόχρονα και επίσης να ε, ενημερώνεται ο κόσμος για τις ε, ε, αλληλεπιδράσεις και οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί να ενημερώνουν και ιδιαίτερα και το οικείο περιβάλλον των ηλικιωμένων γιατί εκείνοι τους δίνουν τα φάρμακα κυρίως, δεν τα παίρνουν μόνοι τους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό και πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσει την έκθεση κατά την άποψή μου είναι ε, η λεγόμενη off-label use. Τι είναι αυτό. Είναι μια χρήση φαρμάκων που συνταγογραφούνται χωρίς να επιτρέπονται για μια συγκεκριμένη εικόνα κλινική. Παράδειγμα, ε, ένα φαρμακό που έχει ε, δοκιμαστεί μόνο σε ενήλικες να συνταγογραφείται σε παιδιά. Δεν επιτρέπεται αυτό. Ή κάτι που ε, είναι ε, κατά των ειδημάτων να το χρησιμοποιεί κανείς κατά των οδυνών το και του. Ή ε, ένα φάρμακο που παίρνεις για την ημικρανία να στο δίνουν μάλλον να το πω αλλιώ, ένα φάρμακο που παίρνει για την επιληψία να στο δίνουν για ημικρανία. Αυτά τα φάρμακα έχουν πάρα πολλέ παρενέργειε για τι οποίε δεν γνωρίζουν τίποτα συχνά οι ασθενεί, γιατί οι γιατροί δεν θέλουν να του κάνουν ενοχλητικέ ερωτήσει οι ασθενεί και βρίσκονται και σε μια γκρίζα ζώνη όταν συνταγογραφούν τέτοια ε, φάρμακα. Υπάρχουν και νομικά προβλήματα όταν δεν επιτρέπεται για μια χρήση να χορηγείται ένα φάρμακο. Αλλά για λόγους κόστους καμιά φορά και πολλές φορές το γράφουν οι γιατροί και μάλιστα αναγκάζονται από τα ασφαλιστικά ταμεία να γράφουν τέτοια φάρμακα. Ε, αυτό δεν επιτρέπεται να συμβαίνει γιατί μπορεί να ενέχει πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους για την υγεία των ασθενών. Άλλο σημείο και τελευταίο. η απέτηση να υπάρχει ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα αποζημιώσεων. Αυτό το βλέπω κάπως επικριτικά. Ας μην το κάνουμε. Αφήστε που το θεωρώ και ανέφικτο, γιατί η πολιτική υγεία και πόσο μάλλον η χρηματοδότησή τη είναι ζήτημα των κρατών μελών. Και βέβαια και στη νομική ερμηνεία προστασία των καταναλωτών υπάρχουν τέτοια ζητήματα και διαφορετική αντίληψη από χώρα σε χώρα. Και το δίκαιό μα δεν έχει εναρμονιστεί. Αφήστε δε που τα συστήματα υγείας διαφέρουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην οργάνωσή τους. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό σύστημα αποζημίωση. Δεν είναι κάτι το υπεύθυνο αυτή τη στιγμή να το ζητάμε και θα κάνω και τροπολογίες για αυτό το θέμα και για τα άλλα που σας προανέφερα. Έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η έκθεση, που είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ τον εισηγητή, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή η έκθεσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζώμερ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετική έκθεση γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο εισηγητής θέλησε να καταλήξει σε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Όλοι μπορεί κάποτε να ασθενήσουμε και είναι απαράδεκτο οι ασθενείς να εκτίθενται χωρίς λόγο σε παραπάνω μολύνσεις. Νομίζω ότι αυτή την εποχή η, διο, αρχίζει να τελειώνει σιγά σιγά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας της σχετικής οδηγίας και μπορεί ο καθένας, πρέπει ο καθένας μάλλον να αποφασίσει τώρα πώς θα επιλέξει που θέλει να τον περιθάλψουν και πώς για την κινητικότητα των ασθενών. Το εδώ το κυριότερο θέμα είναι η ασφάλεια αλλά και η διαφάνεια που πρέπει να επιβάλλουν τα νοσοκομεία για να διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ασφάλεια για τους ασθενείς τους κατά των νοσοκομειακών μολύνσεων. Δυστυχώς δεν συμμετέχα στις, διαπραγματε... στις συζητήσεις αλλά παρακολούθησα τα πράγματα και γι' αυτό κατέθεσα μερικές τροπολογίες, γιατί νομίζω ότι η έκθεση θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένη. Παραδείγματος χάρη να συστήσουμε εθνικές checklist για τα χειρουργία. Αρκεί εδώ να ακολουθήσουμε τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας. Επίσης υπάρχουν διεθνή πρότυπα για την σκανόνες υγιεινής. Αλλά να μην περιοριστούμε στη συλλογή στοιχείων. Αφού πάρουμε τα στοιχεία να τα χρησιμοποιήσουμε ενεργά για να λύσουμε προβλήματα όπου και να βρίσκονται. Είπαν και άλλοι ότι ουσιώδες είναι οι ασθενείς και οι συγγενείς τους να συμμετέχουν ενεργά στην διασφάλιση της ίδιας τους της ασφάλειας. Καμιά φορά το ειδικευμένο προσωπικό δεν αρκεί. Και πρέπει επίσης να μιλήσουμε για τα αντιβιωτικά. Ξέρω ότι το θέμα είναι η ασφάλεια των ασθενών, αλλά για τις μολύνσεις ε, σχετίζεται το θέμα και με τα αντιβιωτικά. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε την πρόκληση αυτή της αντίστασης των βακτηριδίων στα αντιβιωτικά. Και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Σόμερ για το off-label. Συχνά άκουσα να λέγεται να γίνεται λόγος για την χρήση φαρμάκων που δεν στοχεύουν την α ή τη β ασθένεια συγκεκριμένα. Στη Δανία πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε ένα φάρμακο για να προκληθεί το κετός ενώ το φάρμακο αυτό δεν στόχευε ακριβώς αυτόν τον στόχο. Αν λοιπόν χρησιμοποιούνται φάρμακα με στόχο άλλο από εκείνο για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο να γνωρίζει τους κινδύνους δηλαδή. Επίσης Νομίζω ότι η έκθεση θα γίνει αντικείμενο συμφωνίας από όλε τις πολιτικές ομάδες για να ασκηθεί η κατάλληλη πίεση και από τα κράτη-μέλη και σε αυτό μπορεί να συμμετάσχει και η Κομισιόν γιατί σε ενωσιακό επίπεδο μου φαίνεται ότι πρέπει να γίνεται καλύτερα η συλλογή των στοιχείων να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Κορίν Λεπάς εκπροσωπεί το συνάδελφο Τέιλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι θα σας διαβάσω τι μου είπε η συνάδελφος Ρεβέκα Τέιλορ που δυστυχώ δεν μπορεί να προσέλθει σήμερα γιατί έχει ψηφοφορία στην Νομική Επιτροπή ταυτόχρονα για τον Καπινό και μάλιστα στα αγγλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρώση για την πολύ συνοπτική και χρήσιμη έκθεσή του. Ιδιαίτερα νομίζω ότι η έκκλησή του για συγκρίσιμους δείκτες για την ασφάλεια των ασθενών σε ολόκληρη την Ένωση πρέπει να υποστηριχθεί. Επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα την παράγραφο 11 που ζητάει από τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε καλύτερη ταύτιση των υπευθύνων εάν υπάρξει ρήξη στη συνέχεια της αλυσίδας της περίθαλψης. Η παράγραφος αυτή νομίζω ότι θα χρειαζόταν κάποια αποσαφήνιση, δηλαδή για την καλύτερη ταύτιση περιπτώσεων όπου υπήρξε πρόβλημα. Επίσης, Νομίζω ότι χρειάζεται ενδυνάμωση, δηλαδή δημιουργία ενός μηχανισμού αναφοράς των τέτοιων υγειονομικών ατυχημάτων. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία που έχει αυτό το πράγμα. Η παράγραφος 21 και η 35 κάνουν λόγο για ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων του ασθενούς αλλά και τυχόν ατυχημάτων. Τέτοιο επίπεδο προστασίας νομίζω πρέπει να θεωρηθεί ως ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ένωσης. Στην παράγραφο 27 για το σύστημα αποζημιώσεων που πρέπει να εναρμονιστεί σε ενωσιακό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί πολύ πολύ πολύπλοκο στην εφαρμογή του και θα ήθελα περαιτέρω σχόλια του εισηγητή. Υπάρχουν και άλλα θέματα που θα σκεφτώ πριν λήξει η διορία κατάθεσης τροπολογιών και θα έρθω σε επαφή και με ορισμένες υγειονομικές οργανώσεις. Ευχαριστώ πάντως τον κύριο Ρώση για την έκθεσή του, για το σχέδιο έκθεση του. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιανακουδάκη παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μάλλον παντού στην Ευρώπη, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο λέμε ότι όταν υπάρχουν προβλήματα, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ότι πρέπει κανεί να σκεφτεί τι προκλήσει υπάρχουν. Αυτό είναι που συνέχεια γυρνάει στο μυαλό μα, οι προκλήσει. Και αυτό ακριβώ κάνει και η έκθεση, αντιμετωπίζει τι προκλήσει. Ε, θα συμμεριστώ πολλές από τις απόψεις που ανέφερε και ο κύριος Ρώση, ιδίως ότι αφορά τη σημασία να, να ενισχυθεί η ασφάλεια των ασθενών και να προλάβουμε περιστατικά για ασθενείς που βρίσκονται σε νοσηλεία. Στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, η στρατηγική μας για να αντιμετωπίσουμε λοιμώξεις που έχουν να κάνουν με την νοσοκομιακή περίθαλψη, έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά. Πρόσφατα προβλέψαμε μηδενική, πολιτική μηδενικής ανοχής Γι' αυτό καλωσορίζω την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα μας, θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα πρότυπα. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεσης, την παράγραφο 23 της έκθεσης του κυρίου Ρώση, συμφωνώ απολύτως ότι η πρόληψη των λοιμόξεων και νόσων και ο έλεγχος πρέπει να είναι ευθύνη όλων. Όμως θα πιστήσω την προσοχή των συναδέλφων της Επιτροπής μας ώστε να διευκρινίσουμε και τον αριθμό του προσωπικού που θέλουμε ώστε, γιατί δεν είναι ούτε εφικτό ούτε επιθυμητό να δώσουμε συστάσεις για, για την επάντρωση των ε, νοσηλευτικών ιδρυμάτων ακριβώς και λόγω της μεγάλης τους ποικιλία. Η υγειονομική πολιτική εξαρτάται από το πόσο ε, μπορεί να έχουμε και κοινή αρμοδιότητα των κρατών μελών εδώ τα περισσότερα καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές πολιτικές. Οπότε, ε, μια από τις προκλήσεις που προκύπτει εδώ και έχει εντοπίσει ο κύριος Ρώση, είναι το γεγονός ότι τα συστήματα είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους από τη μια χώρα στην άλλη. Συμφωνώ με το σχόλιο σας για την πληροφόρηση των ασθενών. Ωστόσο, αναρωτιέμαι πού θα μας οδηγούσε αυτό, διότι μπορεί οι ασθενείς να φεύγουν πανικόβλητα τα νοσοκομεία και τρέχοντας αν ακούσουν ότι υπάρχει μια λίμωξη ή μπορεί να αρχίσουν να φοβούνται. Ε, πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό με πολύ προσεκτικό τρόπο. Επίσης, μου φαίνεται άστοχο να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα της έκθεσης ιδίας, πρωτοβου... ιδίας πρωτοβουλίας, ώστε να, όπως προτείνει η μπορει να αρχισουν να φοβουνται ε πρεπει λοιπον να γινει αυτο με πολυ προσεκτικο τροπο επισης μου φαινεται αστοχο να χρησιμοποιησουμε τη δυνατοτητα της εκθεσης ιδιας πρωτοβου ωστε να οπως προτεινει η παραγραφος 18, 27 και 37, να δώσουμε στα κάτι μελη να καταλάβουν τι ευθύνε του και πώ θα κατανείμουν τι δαπάνε του. Βέβαια, όμω, μια από τι προκλήσει που αντιμετωπίζει ο κύριο Ρώση είναι πώ θα δοθεί έμφαση στην ε, πρόληψη, λαμβάνοντα υπόψη τα διαφορετικά συστήματα των κρατών μελών και ταυτόχρονα το να πετύχουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Όμω, ε, ανυπομονώ να συνεργαστούμε με τον κύριο Ρώση και να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτή την πρόκληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, η κυρία Κονή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο εξ ονόματος της κυρίας Γκρουστέτ, η οποία μου ζητά να διαβάσω το εξή σχόλιο, το οποίο ε, λέει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθούν διατάξει στην έκθεση ώστε να αντιμετωπιστούν και όσα προκύπτουν από τη χρήση αντιβιωτικών. Θεωρεί αυτή την περίπτωση μια ε, σιωπηρή ε, απειλή η κυρία Γκροστέτ. Η κατανάλωση αντιβιωτικών σε όλα τα κράτη-μέλη εκ νέου ε, παρουσιάζει αύξηση, ιδίω στη Γαλλία. Η κατανάλωση αντιβιωτικών αφορά μάλιστα δικαιολόγια τα περιστατικά και είναι ανησυχητικό να βλέπουμε ότι οι ασθένειε που οφείλονται σε ιού είναι ο πρώτο λόγο συνταγογράφηση αντιβιωτικών. Λοιπόν, αυτή η εξέλιξη είναι θλιβερή διότι ο αριθμός των διαθέσιμων ουσιών έχει μειωθεί περνώντας από 103 σε 84 μέσα σε μια δεκαετία. Η κυρία Γκροστέτ ε, θα προτείνει τροπολογίες για να τονωθεί η έρευνα για την ανακάλυψη νέων αντιβιωτικών και προκειμένου να υπάρξουν δραστικά αντιβιωτικά κατά των παθογενών παραγόντων που έχει αναγνωρίσει και εντοπίσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο των ε, της, των νόσων, της πρόληψης και ελέγχου νόσων του ΕΚΠΕΝ. Θα πρέπει το κέντρο αυτό, όπως λέει και η κυρία Γκροστέτ, να εντοπίσει τους ε, ενδεχομένω θανάσιμους και σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να αποτελούν και μεγάλη απειλή για την δημόσια υγεία γενικότερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Γενική Διεύθυνση της ΣΑΝΚΟ, κυρία Τεστόρη, παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ρώση, ο οποίος αποφάσισε να με κονίσει αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Διότι το θέμα της ασφάλειας των ασθενών, ιδίως στην ε, νοσοκομιακή περίθαλψη, είναι μια από τις προτεραιότητές μας. Ο καθένας από εμά, εφόσον πάει στο νοσοκομείο, έχει 5 10% πιθανότητες να κολλήσει μια λίμωξη. Είναι σαφές λοιπόν ότι πρόκειται για την υπαριθμόν ένα πρόκληση της νοσοκομιακής περίθαλψης. Στην έκθεσή μας και ειδικώ στα συμπεράσματά της συμπίπτουμε κατά πολύ στις απόψεις μας με τον κύριο Ρώση. Ιδιαιτέρως συμμεριζόμαστε την ιδέα ότι εδώ μιλάμε για κοινέ ευθύνες Χρειάζεται να δώσουμε περισσότερη δυνατότητα στους ασθενείς να αναλάβουν την ευθύνη με πληροφόρηση και επίσης με εκπαίδευση και ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού αλλά και την καταγραφή δεδομένων. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση ε, στις ε, νοσοκομιακές Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και θέλουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και επίσης σκεφτόμαστε κατά πόσο χρειάζονται κατευθυντήριε γραμμέ για τα πρότυπα προστασία των ασθενών. Σκοπό μα είναι να υποβάλουμε συστηματικά εκθέσει. Η επόμενη έκθεση για την κατάσταση θα υποβληθεί ε, την επόμενη χρονιά και καλούμε μια από τι επόμενε προεδρίε το θέμα αυτό να το συμπεριλάβει στι προτεραιότητέ τη. Επιπλέον, οι Υπουργοί Υγείας στο προηγούμενο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο συμπεριέλαβαν αυτό το θέμα στις συζητήσεις τους και τα κράτη-μέλη απίθυναν έκκληση ώστε να κουνηθούν κοινέ κατευθυντήριες γραμμές. Ε, λοιπόν, ε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για το θέμα αυτό. Είναι πάντως σημαντικό να ε, διατηρηθεί στην επικαιρότητα. Και απαντώντας την κυρία Οκονή για το θέμα της αντιμοκροβιακής ε, ανθεκτικότητας, κάτι που το παρατηρούμε εδώ και δύο χρόνια, έχουμε εκπονήσει σχετικά πριν από δύο χρόνια πρόγραμμα δράσης και θα συνεργαστούμε με τις αρχές, τις υγειονομικές αρχές, τις κτηνιατρικές επίσης αρχές, ώστε να λάβουμε μέτρα. Είναι κοινό πρόγραμμα δράσης, το οποίο καλύπτει όλους τους αρμόδιους φορεί Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Κύριε Ρώση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που υπάρχει εδώ κοινή ευνοϊκή στάση προς το κείμενο με συνεισφορές ιδιαίτερα θετικές με τις οποίες μπορώ και να συμφωνήσω. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο της Επιτροπής μας και την ε, είδηση, το, την επισήμανση για την αντιμικροβιακή ε, ε, ανθεκτικότητα και την αντίσταση. κάτι που μπορούμε να επιλύ... που αφορά τη χρήση των αντιβιωτικών. Βεβαίω πρέπει εδώ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή εκείνο που κάνει τη συνταγογράφηση ή και ο ασθενή που πολλέ φορέ χρησιμοποιούν εσφαλμένο το αντιβιωτικό. Μια ε, υπό περίπτωση χαρακτηριστική που με μηδενικό κόστο μπορεί να επιληθεί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο φεύγει από το νοσοκομείο και για δυο τρει μέρε ε, παίρνει ένα φάρμακο στο σπίτι του το οποίο του έχει συνταγογραφηθεί. Μπορεί να είναι αντιβιωτικό. την επόμενη μέρα αισθάνεται καλά ο ασθενή, ακόμα και αν έχει συνταγογραφηθεί το αντιβιωτικό μα για 4, 5, 10 μέρε, το παίρνει για 2-3 μέρε και μετά το σταματάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι εκεί ακριβώ δημιουργείται αντίσταση στο αντιβιωτικό. Έτσι, δεν καταφέρνει να φέρει τα, αποτελέσματα του αντιβιωτικού εφόσον ξαναχρησιμοποιηθεί. Εάν φροντίσουμε να ενημερώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο ασθενή και αυτό που φροντίζει τον ασθενή, ε, να είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να επιληφθεί με τρόπο απλό και μηδενικό κόστο. Πάντω, ε, για όσα είπε η κυρία Κονίκ μέρο τη κυρία Γκροστέτ, θα δώσω προσοχή και στο θέμα αυτό των αντιβιωτικών και για όσα είπε η κυρία Γιανακουδάκη, για την ε, κυρία Γιανακουδάκη για το θέμα των προκλήσεων και το πώς πρέπει να δούμε τι γίνεται με νοσοκομεία που έχουν περισσότερα προβλήματα από άλλα, δηλαδή τις διαφορές μεταξύ τους. Λόγω χάρη, εγώ γνωρίζω το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ιταλίας, το Μολυνέτη του Τωρίνο, που είναι και στην περιοχή μου. Εκεί θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα, έχουμε τεράστιο πρόβλημα με ε, από την ε, η οποία έχει να κάνει με τις παλιές υποδομές και την ε, απολύμανση του νερού. Μιλάμε για εκατοντάδες ασθενείς οι οποίοι έχουν επιστρέψει σπίτι τους με αυτή τη λίμωξη. Στις εφημερίδες λοιπόν είδαμε ότι αυτό το θέμα έλαβε μεγάλη δημοσιότητα και τελικά φροντίσαμε να ε, αντιμετωπιστεί η Λεγεωνέλα. Όμως βλέπουμε τι συμβαίνει με τους ασθενείς ε, και τις ε, κακές υποδομές, όπου την προτεραιότητα βεβαίως πρέπει να έχει ο ασθενής και η νοσοκομιακή του ασφάλεια. Για τη μηδενική ανοχή συμφωνούμε απολύτως. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αριθμό προσωπικού στα κράτη-μέλη, ε, αυτό είναι προφανές. Απλώς μπορούμε να απευθύνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη να μην περικόψουν άστοχα τις δαπάνες για τον τομέα της υγείας και όλος ιδιαίτερος για την ασφάλεια των ασθενών. Επίσης στην ε, συνάδελφο Λεπάης που μίλησε εκ μέρους της κυρίας Τέιλορ να την ευχαριστήσω ε, ιδίως για τους συγκρίσιμους δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επειδή όπως είπε και η συνάδελφο Σάλντε Μόζε μας ενδιαφέρει και η διασυνοριακή ε, υγειονομική περίθαλψη. Δεν μιλάμε για έναν Ιταλό ασθενή που θα λάβει περίθαλψη αποκλειστικό στην Ιταλία ή έναν Γάλλο στη Γαλλία αλλά τη δυνατότητα κινητικότητας να ε, κυκλοφορούσαν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και αυτό είναι ένα φαινόμενο ευρύτατο στην Ευρώπη πλέον. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε παρόμοιε συνθήκε ασφαλεία στα νοσοκομεία και να υπάρχει και δυνατότητα ε, διαλογικότητα των συστημάτων μεταξύ του, ώστε να προσφέρουμε ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στου συμπολίτε ασθενεί. Όπω είπε και η κυρία Λεπάζ επίση, όντω για τη βάση δεδομένων μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην, στα πόρτα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, αλλά ε, στην Ευρώπη πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το γλωσσικό ε, θέμα πολλοί ασθενείς μερικές φορές δεν καταφέρουν να συζητήσουν με τον ε, γιατρό που τους φροντίζει ή με το προσωπικό του νοσοκομείου. Ε, η δυνατότητα να υπάρχει μια βάση δεδομένων ε, η οποία θα επιτρέπει να καταλάβει κανείς τι γίνεται με το ιστορικό ενός ασθενή μπορεί να σώσει ζωές. Ναι. Κάποιος ο οποίος είναι άρρωστος μπορεί να μην μπορεί να μου πει σε τι κατάσταση είναι, τι ακριβώ του συμβαίνει. Εάν μπορώ να πάρω ένα χαρτί από τη βάση δεδομένων και να δω ότι έχει αλλεργία στο τάδε αντιβιωτικό ή στο τάδε φαρμακευτικό προϊόν ε, που είναι, χορηγείται στην πήγοντα, προσέχω και δεν του το δίνω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν θέμα και εμπιστευτικότητα η προστασία του ιδιωτικού βίου, αλλά είναι και θέμα τη διασυνοριακή κυκλοφορία των ασθενών. Οπότε πρέπει να προσφέρουμε ασφάλεια στου ασθενεί που πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Εάν δεν είναι σε θέση να μιλήσουν ή να εξηγήσουν, μπορεί εντό εισαγωγικών να πέσουν στην παγίδα ενό οποιοδήποτε σφάλματο. Και κλείνω με την συνάδελφο Σόμερ, την οποία ευχαριστώ, διότι έδωσε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ακόμα και για το ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου προφανώ δεν μπορούμε να έχουμε αποζημίωση ευρωπαϊκή, αυτό είναι σίγουρο, αλλά μπορούμε να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να προβλέψουν όταν υπάρχει σφάλμα ή όταν προκύπτουν προβλήματα ε, ή βλάβε στου ασθενεί του, τότε να, όχι να έχουν την υποχρέωση, αλλά ε, να σκεφτούν την ιδέα να δοθεί αποζημίωση στον ασθενή στο δυνατόν συντομότερα. Μου φαίνεται σωστότερο αυτό και δικαιότερο. Και δυστυχώ σήμερα η οταν προκυπτουν προβληματα η βλαβε του ασθενει του τοτε δυστυχώ είναι ακόμη πολύ στην ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών αποκλειστικά παρά στην ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ όλους και ελπίζω το κείμενο που θα συνταχθεί να, είναι, να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας για όλους προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρώση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 27 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε 12-18 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια δεν έχει ακόμα οριστεί ημερομηνία. Επόμενο θέμα 18 επιστηστική κρίση, περιπτώσει απάτης στην τροφική αλυσίδα και καταπολέμηση αυτών των πρακτικών. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφος Εστέρ Ντελάνγκε η οποία λαμβάνει αμέσω το λόγο. Παρακαλώ κύριε Ντελάνγκε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι πάντε γνωρίζουν ότι η άμεση ε, αφορμή για την έκθεση αυτής της πρωτοβουλίας ήταν υπόθεση με το ε, κρέας αλόγου το οποίο είχε βαφτιστεί βοηθινό, αλλά δεν είναι η μόνη απάτη στα τρόφιμα που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Επίσης, ακόμα και αν φαίνεται, ε, εκ πρώτης όψεως δεν είναι μόνο ζήτημα στο κρέας. Τα τελευταία χρόνια ε, είχαμε δει σε ψωμί αλάτι που ήταν για τους δρόμους, για τα χιόνια, όχι βρόσιμο αλάτι, ακόμα και αυγά ε, βαφτίστηκαν βιολογικά που σίγουρα δεν ήταν σε καμία περίπτωση βιολογικά. Και την τελευταία διετία περίπου έχουμε δει και άλλες τέτοιες απάτες στα τρόφιμα. Είναι ευρύτατα διαδεδομένο το πρόβλημα. Προχτές κάναμε ακρόαση για αυτό το ζήτημα και τι προέκυψε ως συμπέρασμα. Ε, ότι έχει έρθει η ώρα επιτέλους να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να γράψουμε την έκθεση πρωτοβουλίας. Διότι, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, σε αντίθεση με την Αμερική, δεν έχουμε καν ορισμό τι εστία απάτη στα τρόφιμα. Ε, ο καθένας σκέφτεται διάφορα πράγματα νοθείας, αλλά δεν υπάρχει στην Ένωση ενιαίος ορισμός. Κατά την άποψή μου ε, θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτόν τον ορισμό διάφορα στοιχεία. Πρώτον, ο δόλος και ε, ο στόχος, το οικονομικό όφελος. Αυτά τα δύο έχουν σχέση μεταξύ τους. Δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν νομίζω. Είναι πραγματικά εσκεμμένο ε, με δόλο, ε, με στόχο το οικονομικό συμφέρον. Είναι σχορκέρδια το αποτέλεσμα μπορεί να είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, αλλά όχι απαραίτητο. Ε, δεν σημαίνει ότι έχει, πάντα υγειονομικό κίνδυνο. Ε, συμβαίνει το εξής πολλές φορές. Ε, κλονίζεται ο κόσμος στην εμπιστοσύνη του που έχει στα τρόφιμα και αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό για να μας απασχολήσει. Κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα παράδοξο, γιατί κάθε επιστημονική μελέτη δείχνει ότι ουδέποτε ήταν τόσο ασφαλή τα τρόφιμά μα. Ε, παρά αυτά ο κόσμο δεν εμπιστεύεται τώρα όταν τον τουζείζουμε τέτοια πράγματα σε μια ετικέτα μάλιστα που είναι και ευρωπαϊκή και την ε, επισημαίνουμε και λέμε εμεί τι πρέπει να γράφει, ο κόσμος δεν την εμπιστεύεται. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να βασιζόμαστε στην ασφάλεια των τροφίμων και ε, ε, η απάτη όμως είναι πολύ ευρύτερη από την ασφάλεια. Το νομοθετικό πλαίσιό μας ε, είναι πάρα πολύ προσανατολισμένο στην επισήμαση, στις ετικέτες. Για το general food ας πούμε αυτό μας ενδιαφέρει είναι η ετικέτα να μην είναι παραπλανητική. Αυτές είναι οι λαβές που έχουμε για να ε, αντιμετωπίσουμε την απάτη στα τρόφιμα. Αρκεί όμως ε, για να αντιμετωπιστεί αυτή η νοθήνα. Αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξει το πλαίσιο έτσι ώστε ε, να υπάρχει ένας ορισμός για να μπορούμε να ανοιχνεύουμε καλύτερα και να αντιμετωπίζουμε αυτές τις απάτες. Μια σειρά στοιχείων λοιπόν που κατά την άποψή μου ανήκουν σε αυτό, το πλαίσιο έτσι που χρειάζεται για να το εξασφαλίσουμε, είναι το θέμα της ανάλυσης κινδύνου, του ρίσκου, δηλαδή πώς θα καταλάβεις ποιες εταιρείες πρέπει να παρακολουθείς και να ελέγχεις. Ας πούμε, στο κρέας μπορεί κάποιος ε, να κάνει κρεοσκοπικό έλεγχο σε ένα σφαγείο, να ε, περνάνε από μπροστά του σφάγια όλη μέρα σε μια αλυσίδα και να είναι εντάξει. Αλλά στην Ολλανδία, ε, σε αυτή την εταιρεία που κατηγορείται, δεν έχει πατήσει ποτέ κανείς για έλεγχο. Γιατί ο έλεγχος γίνεται στα σφαγεία, ο κρεοσκοπικός, αλλά δεν πάει κανείς στον έμπορο να δει τι πουλάει και τι αγοράζει. Θα πρέπει λοιπόν να γίνονται οι έλεγχοι εκεί που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για νοθεία και απάτη. Επίσης χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενεχομένων. Στην Ιρλανδία υπάρχει το γραφείο ε, για τα τρόφιμα και τα κτηνιατρικά Food and Veterinary Office ε, και ε, έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να υπάρχει ένα διαβατήριο για τα υποειδή. Είναι γνωστά αυτά και το, βόιο, και το ήπιο κρέας, συγγνώμη, το κρέας αλόγου δηλαδή πώς κυκλοφορεί στην αγορά ε, αυτό επίσης παρακολουθείτε. Είναι ένας τομέας που πρέπει να ελέγχεται. Δεν έχει συμβεί όμως αυτό. Και επίσης η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρατών Μελών είναι πολύ σημαντική και μας ενδιαφέρει. Παράδειγμα, κοιτάξτε το σκάνδαλο στην Ιρλανδία. Τρεις εταιρείες οι Ιρλανδοί δεν μπορούν να τη συλλάβουν γιατί η και απάτη έχει γίνει εκτό Ιρλανδίας. Έχουν δώσει την ενημέρωση μεν, αλλά δεν ξέρουμε αν διώχθηκαν και τι συνέχεια δόθηκε. Γι' αυτό χρειάζεται διακρατική συνεργασία. Επίση, είναι ενδιαφέρουσα ιδέα αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε ε, το σύστημα που υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για τα τρόφιμα και τι ζωοτροφές να ε, το επεκτείνουν και για την απάτη. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη χρησιμότητα αυτό, γιατί το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση τι είναι, απλούστατα μια βάση δεδομένων για ανταλλαγή πληροφοριών. Ότι κάποια στιγμή υπάρχει μια κρίση και να ενημερωθούν τα κράτη γρήγορα ότι κάτι προέκυψε. Ε, χρειάζεται όμω εκεί να υπάρχει και η δυνατότητα ανάλυση, όχι απλώ να υπάρχουν στοιχεία που να κυκλοφορούν, αλλά να τα αναλύουν και να βγάζουν και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Κυρώσεις επίσης είναι κάτι που θα πρέπει να μα απασχολήσει. Προσοχή όμως διότι η αρμοδιότητα παραμένει εθνική. Να σας δώσω και πάλι το παράδειγμα το Ιρλανδικό. Κατάφεραν οι Ιρλανδοί να βρουν ποια ήταν η εταιρεία που έκανε την απάτη. Σε Ιρλανδικό έδαφος. Και διώκεται ε, ποινικά. Αν το καταφέρουν αυτό, το μέγιστο ε, κέρδος ε, είναι 30.000 ευρώ από το πρόστιμο, ενώ ένα και μόνο κοντέινερ με το λάθος κρέας αποφέρει κέρδος 65.000. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το οικονομικό κίνητρο και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί κάπως στα πρόστιμα και τις κυρώσεις από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, μητρό εμπόρων, καταγραφή, να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Ιδιαίτερα όταν επεξεργάζονται στη συνέχεια το προϊόν αυτή, το αποσυσκευάζουν, το επανασυσκευάζουν και κάνουν διάφορους χειρισμούς, ε, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τι να ζητήσουμε από την έκθεση και περιμένω και από τους συναδέλφους ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι ο ορισμός που να ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην Ευρώπη, υπάρχουν κάποιες τάσεις ε, για απάτες τροφίμων, ποια είναι τα υποκείμενα αίτια, αλλά κυρίως ποια είναι τα διδάγματα που μπορούμε να εξαγάγουμε για το μέλλον. Έχω και μια σειρά από στοιχεία εδώ που πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στην έκθεση, αλλά κυρίως περιμένω με ενδιαφέρον και περιέργεια να ακούσω τους συναδέλφους. Ε, θα ακολουθήσει η συγγραφή του έργου. Πριν φύγω για διακοπές, περίπου τέλη Ιουλίου να περιμένετε ένα σχέδιο έκθεση από πλευρά μου για τη μετάφραση έτοιμο έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε το Σεπτέμβριο. Αλλά προς το παρόν αυτό που με ενδιαφέρει να ακούσω τους συναδέλφους. Να ακούσω τις ανησυχίες, τα μελήματα αλλά και τις επιθυμίες τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Εστέρ. Η Κορίν ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την συγγήτρια αλλά και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες που κάνουν τη δουλειά τους με όλο και λιγότερα μέσα και απεκάλυψαν αυτή την απάτη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι την περίπτωση του αλογίσκου κρέατος δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε σαν μια ατομική απάτη που δεν μας αφορά. Υπάρχει εδώ ένα συλλογικό λάθος. Λένε ότι έχουμε την καλύτερη νομοθεσία του κόσμου. Ναι, στα χαρτιά, αλλά δεν υπάρχει έλεγχος. Και υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί που επιτρέπουν την απάτη. Έχουμε και εμείς λοιπόν ένα μερίδιο ευθύνης γιατί αντιταχθήκαμε στη σαφέστερη σήμανση για την καλύτερη προοφορήση των καταναλωτών. Επίσης δεν θελήσαμε να επιβληθεί έλεγχος όσων συσκευάζουν τα τρόφιμα. Όλες οι υγειονομικές και υπηρεσίες και εκείνες που αφορούν τα τρόφιμα πρέπει να ελέγχονται. Παραδείγματο χάρη είναι αυτά που κάνει η γαλλική Εύσα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λοιπόν δεν έλεγξαν καλά την σφαγή των αλόγων σε κοινοτικό επίπεδο, ούτε τις ενδείξεις που υπήρχαν και έτσι υπερβολικά αργά αποκαλύφθηκαν όλα. Εδώ πρόκειται για έλλειψη στη λειτουργία του όλου οικονομικού συστήματος. Οι κρίσεις και οι απάτες δεν αφορούν μόνο το κρέας αλόγου, αλλά και άλλους τομείς όπως παραδείγματο χάρη την ανακάλυψη απαγορευμένου γενετικά τροποποιημένου σύτου. Η οδηγία λοιπόν 178-2002 πρέπει να εφαρμοστεί για τη διοίκηση της κοινοτικής υπηρεσίας ελέγχου. για να αποφευχθεί μια προσεχής κρίση της οποίας δεν γνωρίζουμε καν το αντικείμενο και τους υγειονομικούς κινδύνους, ούτε την επίπτωση που θα έχει στην αξιοπιστία των καταναλωτών, πρέπει η Κομισιόν συστηματικά να κάνει ελέγχους DNA και για όλες τις πρωτεΐνες που μπαίνουν στην διατροφική αλυσίδα. Ευχαριστώ. Για το θέμα αυτό που είναι τόσο σημαντικό και που ξεπερνάει τα καθαρά διατροφικά. Γίνεται πολιτικό γιατί η εμπιστοσύνη μη των καταναλωτών είναι θέμα καθημερινής ζωής και του ελέγχου που είμαστε ή δεν είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε στα τρόφιμα. Ευχαριστώ. Ο Μπαρτ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ με την εισαγωγή της ε, Λάγκε. Είναι πραγματικά πολύ πλήρης η απεικόνηση και η σχεδιαγράφηση του προβλήματος. Είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε ε, ε, και θα συνεργαστούμε καλά, είμαι βέβαιος. Πραγματικά είναι κρίσιμο το θέμα του ορισμού. Χρειάζεται ένα πολύ καλός ορισμός για την απάτη και την οθεία στα τρόφιμα και ε, αυτά τα δύο στοιχεία που προτείνει η Εστέρ είναι πολύ καλά. ο δηλαδή ο δόλος και το οικονομικό συμφέρον και όφελος. Τα κράτη-μέλη καλούνται να παίξουν ένα κρίσιμο ρόλο, πρωταγωνιστικό στην καταπολέμηση ε, της απάτης, γιατί συχνά είναι διεθνή τα δίκτυα και περίπλοκα και ε, όσο πιο περίπλοκο είναι, ε, πιο, τόσο πιο εύκολη γίνεται η νοθεία. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ε, πρέπει να σας πω, δεν ήμουν παρόν προχτές ε, στην ακρόαση γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού αλλά έστειλα του βοηθό μου και με ενημέρωσε πάρα πολύ καλά και ακούω ότι ο κύριος Κουντελέ μίλησε πολύ καλά για το σύστημα αυτό έγκαιρης προειδοποίησης και εξήγηλε ότι ίσως να το ξαναδούμε, να το αναθεωρήσουμε και να το αλλάξουμε και να συμπεριλάβει και την ασφάλεια τροφίμων και να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου της απάτης στα τρόφιμα. Υπάρχει τεχνογνωσία στα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου και στη χρήση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και προς την κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως, όπως είπε και η Εστέρ, αυτά συμβαίνουν κατόπιν εορτής. Μόλις ξεσπάσει ένα σκάνδαλο και το ανακαλύψεις, αλλά μη τι άλλο να κοινοποιείται γρήγορα. Ναι στον έλεγχο, ναι στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι απολύτως απαραίτητο, ιδιαίτερα στις συνοριακές παραμεθόριες περιοχέ και όταν πρόκειται για διεθνείς πύρες. Ε, τώρα τα πρόστιμα και κυρώσεις είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα, διότι το είπε και η Έστερ αυτό, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα πρέπει να δούμε την αναλογικότητα κάπως των προστήμων, έτσι να έχουμε περίπου παρόμοιες κυρώσεις. Ε, το ε, είχα υπόψη μου αυτό. Ασχολήθηκα πάρα πολύ καιρό ε, με τους αυξητικούς παράγοντες ε, στην κτηνοτροφία. Ε, δεν φοβούνται να κάνουν διάφορες κομπίνες ή κακοποιοί γιατί το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ ενώ το κέρδος πολλαπλάσιο. Η λασιμότητα επίσης πώς μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα, αλλά και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ο οργανισμός της Ιρλανδίας, το Γραφείο Κτηνιατρικών και Τροφίμων. Κάνουν καταπληκτική δουλειά εκεί οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη διαφάνεια. Ε, κοιτάξτε στην ιστοσελίδα του σας το συνιστώ, είναι πάρα πολύ καλή, το είπε και η Έστερ και ε, με το κρέας αλόγου το χειρίστηκαν πάρα πολύ καλά. Ε, έκαναν πολύ καλή ενημέρωση και αν όλα αυτά που είχαν συστήσει στο παρελθόν ε, τα είχαμε ακολουθήσει, ίσως να αποφεύγαμε τέτοιες καταστάσεις. Και θέλω να επενέσω αυτό το γραφείο και θα πρέπει ε, εδώ στην Επιτροπή μας, στο Κοινοβούλιο, να ζητάμε ενδεχομένως να διοργανώνεται ετησίως μια συζήτηση μια ανταλλαγή απόψεων με τους ανθρώπους από το γραφείο αυτό, από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, ενδεχομένως και με τον αρμόδιο επίτροπο και να πούμε. Τα πεπραγμένα, ε, το γραφείο κτηνιατρικών και τροφίμων αντιμετώπισε αυτά τα μεγάλα προβλήματα, αυτά ήταν οι γραμμές. Υπάρχει προβληματικό τομέα όπως είναι το κρέας αλογού ή κάτι άλλο. Υπάρχουν χώρες που πραγματικά δεν είναι καλή η έλεγχη. Και έτσι σε τίσια βάση να κάνουμε ε, και ένα, αυτό που λένε στα αγγλικά naming and shaming, ε, δημοσίευση και διαπόμπευση των ονομάτων ορισμένων ε, που παρανομούν και στα κράτη-μέλη επίσης αναχώρα μπορούμε να συστήσουμε να γίνουν στις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές τους επιτροπές. Θα ήταν φανταστικό για μένα στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή κάθε φορά να γίνεται μια ετήσια ε, παρουσίαση. Ας πούμε στο Βέλγιο το 12 έκανε πέντε επιθεωρήσεις το ε, κτηνιατρικό γραφείο και ε, τροφίμων και έκανε συστάσεις. Τι έγινε στη συνέχεια, πώς εφαρμόστηκαν αυτά από τις κτηνιατρικές αρχές, από τις αρχές δημόσιας υγείας, από το Υπουργείο Γεωργίας, ξέρω εγώ, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να αναβαθμίσουμε και πολιτικά τη δουλειά αυτού του οργανισμού και να προλαμβάνουμε και κακές καταστάσεις. Τέλος, ε, με τον α ή β τρόπο θα πρέπει κάπως να οργανώσουμε την τροφική ε, λυσίδα. Το είπε και η Έστερ, ε, θα το ξαναπεί φαντάζομαι. όσο πιο περίπλοκη είναι η τροφική αλυσίδα, όσο πιο μεγάλα ταξίδια κάνουν τα τρόφιμα από τη μια χώρα στην άλλη, τόσο πιο εύκολο είναι να νοθευτούν και να εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Αυτό είναι και το πρόβλημα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πολύ σύντομες ε, τροφικές αλυσίδες. Αυτό έχει και πλέον ε, γενικότερα. Όχι μόνο ότι οι άνθρωποι που κάνουν εμπόριο μεταξύ τους γνωρίζονται καταρχήν, αλλά ε, είναι πολύ μεγαλύτεροι και οι δεσμοί μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Είναι μικρές οι αποστάσεις που διανύουν τα τρόφιμα και πολύ καλύτερη η αγορά. Άκουσα την Τρίτη ε, ότι στην ακρόαση υπόθηκε ότι ε, όλη αυτή η ιστορία με την ετικέτα και την προέλευση δεν καταπολεμά την απάτη. Δηλαδή δεν είναι μέσω καταπολέμησης απάτης αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μελέτες αντικτύπου και ε, θα κάνει και πρόταση το φθινόπωρο για να διευρεθεί το σύστημα για το βόλιο κρέας και την προέλευση και την ετικέτα. Αυτή τη στιγμή ανακαλυφθεί μια απάτη, βοηθάει και η ετικέτα για να καταπολεμηθεί αυτή η νοθεία. Αλλά όταν ε, ε, υπάρχει και πλαστογραφία των εγγράφων δεν είναι εύκολο να καταπολεμηθεί, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτές ορισμένες πρώτες σκέψεις ε, και θα έχουμε την ευκαιρία και το χρόνο να ανταλλάξουμε απόψεις επί της ουσίας περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Γκέρλι. Ευχαριστώ. Τα περισσότερα από ήθελα να πω ήδη υπόθηκαν, οπότε δεν θέλω να σας καθυστερήσω, απλώς μια-δυο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Εστέρη για την ακρόαση, την οποία μπόρεσα να συμμετάσχω εν μέρη. Όσα δεν άκουσα, ε, τα διάβασα και είδα ότι ήταν ε, πολύ ενδιαφέροντα όσα υπόθηκαν, όσο ό,τι αφορά τι απειλέ που δεν το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο με το κρέα αλόγου, όπω ονομάστηκε, δεν έχουμε τις πληροφορίες τελικά που πιστεύαμε ότι πρέπει να έχουμε. Αυτό φάνηκε. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρουμε και πώς να τις βρούμε. Είναι... Ήταν μια χαρακτηριστική υπόθεση, μας έδειξε πώς λειτουργεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, πώς θα έπρεπε να λειτουργεί και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί. Οι γενικές μου παρατηρήσεις είναι ότι έχοντας μελετήσει το θέμα αυτό, με αρκετή προσοχή, δεν είμαι βέβαιη ότι πρέπει να προτείνουμε νέα νομοθεσία. Διστάζω βέβαια να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, θα έπρεπε ίσως να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός. Δεν εννοώ ένας κανονικός ευρωπαϊκός οργανισμός, κάποιο είδους φορέας, μια ε, βασική επιτροπή, ε, ένα σημείο συνάντησης που συστηματικά ε, να συγκεντρώνει δεδομένα και να τα δημοσιεύει για τέτοια στοιχεία όπως οι δοκιμές διότι αληθεύει ότι με το σχέδιο των πέντε σημείων που έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ένα διεξοδικό πρόγραμμα δοκιμών. Θέλουμε όμως αυτό να γίνεται συστηματικά και κυρίως ε, σε μια βάση διαφάνειας. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχουμε κάποια παρακολούθηση του όλου θέματος, εάν όχι επιρροή στο πώς θα λειτουργεί, αλλά τουλάχιστον κάποια παρακολούθηση, ώστε να, είμαστε, να ενημερωνόμαστε τακτικά. Εάν γινόταν αυτό που θα ήταν και μια ενεργό συμμετοχή στο όλο, στο όλο θέμα, αυτό θα εξυπηρετούσε και τα κρατημέλη και τους ε, ε, μας που χρειάζονται κάτι τέτοιο και δεν θα το αφήναμε τελείω στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν λέω ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμω δεν είναι αρκετά διαφανή αυτή η δουλειά, ούτε αρκετά ανοιχτή για το κοινό, ούτε ε, καθησυχάζει αρκετά το κοινό. Και είναι σημαντικό γιατί κάποιοι μιλάνε για περισσότερου κανόνε, περισσότερη νομοθεσία. Εγώ πιστεύω ότι αυτή θα ήταν λάθο προσέγγιση. Α αξιοποιήσουμε όσα διαθέτουμε ήδη. Αλλά τουλάχιστον να έχουν ευκολότερη πρόσβαση οι πολίτε. Πραγματικά το θέμα που επανειλημμένω ανέφερε η Εστέρ πρέπει να το δούμε με προσοχή. Αυτό που ανέφερε στην ακρόαση, τη διασυνοριακή συνεργασία. Αυτό δεν έχει διερευνηθεί όσο του αξίζει. Θα πρέπει να έχουμε ένα, μια λυσίδα διαφανή και σαφή, ώστε να ξέρουμε πώς μπορούμε να εργαστούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Άντερσον εκπροσωπεί σήμερα η καρτή Καλλιωτάρ. Παρακαλώ. Με ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος της Μαρτίνα Άντερσον, δυστυχώς κολλείεται και απουσιάζει σήμερα και ε, θα την ε, αντικαταστήσω εγώ. Θέλει και εγώ φυσικά να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα την κυρία Ντελάνγκε και για την εισαγωγή της, γιατί πραγματικά εντόπισε τον πυρήνα των πραγμάτων και τα περιέγραψε πολύ ωραία, αλλά και για το ατελιέ, την ακρόαση που έγινε την περασμένη Τρίτη, ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική αυτή και ενημερωτική. Και όπως υπόθηκε ήδη, μιλήσαμε πολύ για το ε, κρέας αλόγου και το σκάνδαλο και αν πρόκειται για θέμα ασφάλειας των τροφίμων ή, θέμα απάτης και νοθείας στα τρόφιμα, ό,τι και να είναι, δεν επιτρέπεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και ως συνομοθέτης εμείς έχουμε ρόλο. Θα πρέπει ο καταναλωτής ε, να γνωρίζει τι τρώει. Έχει το δικαίωμα. Θα πρέπει να ενημερώνεται, αλλά όχι μόνο. Αν δεν αντιμετωπίζεται εγκαίρως η απάτη στα τρόφιμα μπορεί ε, να σημάνει και πρόβλημα στην ασφάλεια των τροφίμων και ε, να είναι ο κίνδυνος πολύ μεγαλύτερος από ένα οικονομικό κίνδυνο. Και θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Ε, και ο κύριος Πουντλέ ήταν επίσης παρόν στο ατελιέ αυτό, στο εργαστήρι, μίλησε για ένα πρόγραμμα δράσης πέντε σημείων του Επιτρόπου Μπόρτς. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται πάντα σε αυτά τα θέματα, αλλά θα ήθελα καλύτερα να δω νομοθεσία ή αν όχι καινούργια, προσαρμογή παλιάς ε, ε, νομοθεσίας για να έχουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά το πρόβλημα. Επίσης, ε, ακούστηκε και προηγουμένως ότι σήμερα δεν υπάρχει ορισμός για την απάτη στα τρόφιμα. Συμφωνώ με τα δύο στοιχεία, το δόλο και το οικονομικό όφελος και θα πρέπει να τα γράψουμε και μάλιστα να μιλήσουμε και για τη δόλια απόκρυψη στοιχείων, όχι μόνο παραπληροφόρηση. Επίσης, οι διάφοροι ζωέμποροι και έμποροι κρεάτων θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά, να αναγράφονται σε ένα μητρό και να έχουν υποχρέωση κοινοποίησης. Δηλαδή όταν είσαι εμπορο και διακινείς κρέα και δεν σε λέει το μητρό να απαγορεύεται ε, και να μην έχουν δυνατότητα ε, εμπλοκή σε αυτό το εμπόριο διάφοροι άσχετοι παράγοντες. Σε ό,τι αφορά τώρα το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, καλό θα ήταν να διευρυνθεί αυτό και ε, να καλύπτει και την οθεία στα τρόφιμα. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό, αλλά μάλλον από σπασματικά και χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Εγώ θα πρότεινα να το ε, διευρύνουμε και να καλύπτει και την απάτη στα τρόφιμα έτσι ώστε ε, οι αρμόδιες αρχές, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούν να επεμβαίνουν ε, στεναρότερα. Επίσης γνωρίζω ότι διώκονται ποινικά οι υπεύθυνοι αλλά είναι ζήτημα των κρατών μελών αυτό Ε, θα πρέπει να είναι τα πρόστιμα τέτοια και οι κυρώσεις ώστε να δρουν ε, ε, αποτρεπτικά, αλλά αυτό να το επομίζονται τα κράτη-μέλη. Να πω και δύο λόγια για την ετικέτα, για τη σήμανση της προέλευσης. Είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για να έχει περισσότερες πληροφορίες ο καταναλωτής για το προϊόν και όσο καλύτερα ενημέρωση είναι ο καταναλωτής, τόσο λιγότερο κινδυνεύει να παραπλανηθεί και ιδιαίτερα για το κρέας θα πρέπει οπωσδήποτε να γραφτεί προέλευση. Κοιτάξτε τι έγινε με τα λαζάνια και το κρέας αλόγου. Ε, θέλω οπωσδήποτε να το τονίσω αυτό, την ετικέτα του, της χώρας προέλευσης. Και όχι μόνο σε αυτή την νομοθεσία, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πολύ περισσότερο η νοθεία στα τρόφιμα και η απάτη αυτή και προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε με την Επιτροπή αυτή ε, μία έκθεση για τη σήμανση του βοήου κρέατος. Θα πρέπει να ε, τηρήσουμε τις θέσεις που είχαμε στο παρελθόν για την κλωνοποίηση, γιατί και τέτοια θέματα ε, είναι ευαίσθητα, είναι επιρρεπή στην απάτη και αν κάνουμε σε αυτή την έκθεση, ε, αν αναφέρουμε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θέμα, δεν θα μπορέσει να τα χωρέσει η έκθεση. Ευχαριστώ. Εδώ κλείνει ο κατάλογος των σκιωδών εισηγητών και αρχίζει να πιέζει ο χρόνος. Ε, παρακαλώ τους υπολείπους ομιλητές, ο Κονή, Ρώση και Σόμερ, να περιοριστούν στο 1,5 λεπτό έκαστος η Σοφία Οκονή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σήμανση του βοήου κρέατος είναι κάτι που μας συνδέει εδώ και μερικούς μήνες κύριε Πρόεδρε γιατί εγώ είμαι συγγήτρια για αυτό το θέμα και άκουσα το μήνυμα της κυρίας Λιωτάρ και σκεφτώ το αναλύουμε τώρα και θα συνεργαστούμε και για τα κλονισμένα με ωμέγα ζώα, κλωνοποιημένα. Από αυτά που μας αναφέρατε βλέπω ότι με το πολλά συμφωνώ. Το πρόβλημα δεν είναι δημόσια υγεία αυτό το πράγμα του σκανδάλου που αναφέρεται. Αλλά είναι θέμα ποιότητας και δεν υπάρχει αρκετός έλεγχος. Ούτε κυρώσεις. Σας υπενθυμίζω ότι στη Γαλλία μία μητέρα που κλέβει ένα μπιφτέκι σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν είναι η πρώτη φορά, τότε τιμωρείται αυστηρότερα από την εταιρεία που εξαπάτησε όλο τον κόσμο στη Γαλλία. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι στον έλεγχο της ποιότητας των κρεάτων, αλλά και στις κυρώσεις. Ε, ε, l'autocontrôle Euh, euh. Λοιπόν, το βασικό πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Υπάρχει ας πούμε το σκάνδαλο πολλών θεμάτων, όχι μόνο στο κρέας και σε άλλα και πρέπει να μπορέσουμε να επιβάλλουμε ένα πλαίσιο για τους ποιοτικούς αυτούς ελέγχους. Και επίσης να σκεφτούμε το θέμα των εμπόρων και των τρέιντερς τροφίμων. Τα προετοιμασμένα φαγητά α, καθώς και τα μέταλλα που μπορεί να περιέχουν. Και τις μαζικές πωλήσει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας κώδικς ποιότητας για αυτές τις μαζικές πωλήσει. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είναι δύσκολο αυτό το θέμα, πραγματικά περίπλοκο, ευρύτατο και αφορά πολλά συμφέροντα και πολλούς Ευρωπαίους καταναλωτές. Στον τίτλο γίνεται λόγος και για την επισητιστική κρίση. Αυτό τι σημαίνει. Θα συζητήσετε επίσης και με το πώς μπορούν να επανακτηθούν αυτά τα τρόφιμα που έχουν κατασκευθεί και καταλήγουν στα απορρίμματα. Υπάρχει το θέμα της ετικέτας και το made in της προέλευσης. Σήμερα μπορεί ο καθένας να εισάγει προϊόντα που έχουν παραχθεί στο εξωτερικό, να το, όπως συσκευάσει στην Ιταλία να βάλει νέα συσκευασία και να γράφει Made in Italy. Και εσείς πού θα βρείτε ε, από πού έχει εισαχθεί το προϊόν και πόσο μάλλον ο τελικός καταναλωτής. Μια σαφής ετικέτα επίσης επιτρέπει στους πολίτες και στους καταναλωτές να γνωρίζουν τι ακριβώς καταναλώνουν. Προσωπικά πήγα και είδα ακριβώς τι σημαίνει γεύση φράουλα. Ε, πήγα και το ψάξα αυτό. Είναι χημικές ουσίες, 50 παρακαλώ, συγκεντρωμένες ε, και στην ετικέτα τη γράφει άρωμα, φράουλας, ενώ είναι 50 ουσίες. Άρα, παίρνει μια τσίχλα και τη μασάς και νομίζεις ότι είναι μαστίχα φυσική, καθόλου. Οι τσίχλες ε, σήμερα είναι 99% πετρέλαιο. Δεν το ξέρουμε όταν μασάμε τσίκλα και ο Ευρωπαίος καταναλωτής ακόμα λιγότερο. Η κυρία Ζώμα. Ναι. Χαρά που θα κάνει ο καταναλωτής άμα ε, έχει και όλα τα συστατικά, τα γράφει ετικέτα, πόσα αρώματα έχει τα 50 μέσα, δεν θα υπάρχει συσκευασία. Ε, αγαπητή κυρία Λεωτάρ, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ο κανονισμός για την ενημέρωση για τα τρόφιμα ε, είναι στη φάση της υλοποίησης και ε, ελέγχεται η προέλευση των κρεάτων και η ετικέτα. Τώρα να ζητάμε πιο αυστηρέ ετικέτες για κάτι ε, που έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό το θεωρώ υπερβολικό. Συμφωνώ μάλλον με την κυρία Γκέρλινγκ που ζητεί να εφαρμόσουμε την κείμενη νομοθεσία για τα τρόφιμα. Δεν μπορούμε συνεχώς να βγάζουμε νέους ε, νόμους. Η απάτη δεν θα σταματήσει να υπάρχει, ό,τι νόμο και να έχεις. Ο απατεώνας την ετικέτα απλά στο γραφεί. Ό,τι και να του επιβάλλει η ετικέτα και έχουμε την οθεία και το σκάνδαλο μετά και την απάτη. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτά τα θέματα είναι το εξής. Θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη το ποινικό δίκαιο να το εναρμονίσουν. Δεν επιτρέπεται σε μια χώρα κάποιος που κάνει τέτοια απάτη και νοθεύει ένα τρόφιμο να τιμωρείται υποδειγματικά και σε άλλη χώρα του στέλνουν ε, μία επίπληξη γραπτή και πεθαίνει από τα γέλια στη συνέχεια. Και δεν αρκούν επίση τα χρηματικά πρόστιμα, θα πρέπει να είναι ψηλά πρόστιμα, οι ποινές φυλάκισης. Μόνο έτσι ε, ε, εδρά αυτό αποτρεπτικά, όταν όλο φοβάται ότι θα πάει φυλακή. Κατά τα άλλα, θεωρώ θαυμάσια την έκθεση, καταπληκτική αγαπητή Εστέρ. Και τώρα προσζητώ συγγνώμη γιατί εδώ και μισή ώρα έπρεπε να είμαι σε ένα άλλο ραντεβού που είχα. Και πέρασε και το χρόνο αγόρευσή σου, κατά τα άλλα. Λοιπόν, <laughs> τελειώσαμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Τεστόρη, νομίζω. Ξενόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. This is my expert, my expert here on the fraud. Εδώ ο ειδικό μου περιαπάτης θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε είναι δύσκολο να αντικαταστήσει την κυρία Τεστόρη γιατί είναι πολύ, έχει μεγάλο πάθος. Θα ήθελα να σας πω κυρία Ντελάνγκ ότι συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτές σας τις ανησυχίες. Η έκθεση είναι πολύ επίκαιρη διότι εδώ και 15 χρόνια διαπιστώνουμε απάτες στα τρόφιμα σε μεγάλη κλίμακα. Δυστυχώς η αντίδρασή μας ήταν αρκετά περιορισμένη μέχρι τώρα, αλλά ο Επίτροπος Μπόρτς κατάλαβε τι σημαίνουν επιτέλους όλα αυτά με το τελευταίο σκάνδαλο για το κρέας και όπως ξέρετε ε, θέλει να εφαρμόσει ένα σχέδιο σε πέντε σημεία το οποίο έχετε, είχατε την ευκαιρία να το συζητήσετε με εκείνον. Τώρα για τον ορισμό της απάτης υπάρχει νομικό πρόβλημα, δεν έχουμε τέτοιο ορισμό στο General Food Law προβλέπεται σε ένα άρθρο ότι ο στόχος της νομοθεσίας για τα τρόφιμα είναι να αποτραπούν οι απάτες για τα τρόφιμα καθώς και κάθε πρακτική που μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε λάθος, ε? Δεν είναι πραγματικός ορισμός της απάτης, αλλά είναι μια κάποια νομική βάση που επιτρέπει την ε, καταπολέμησή της. Και βέβαια συμμεριζόμαστε και τη θέση της κυρίας Ντελάνγκ ως προς τις δύο έννοιες πρόθεση και κέρδος. Θα θυμάστε με την Εσκερίκη Ακόλη που προερχόταν τελικά από την Αίγυπτο και παρόλα αυτά προκάλεσε το θάνατο 55 ανθρώπων χωρίς να πρόκειται για απάτη. Ήταν απάτη μόνο ως προς τη σήμανση αλλά όχι ως προς την υγεία το θέμα του αλογίσιου κρέατος. Γιατί η ετικέτα ανέφερε βόλιο κρέας, το οποίο είναι τρεις φορές ακριβότερο από το αλογίσιο. Υπάρχει λοιπόν εκεί η έννοια του κέρδους. Τώρα εξετάζουμε πώς να δημιουργήσουμε ένα νομικό υπόβαθρο για τον ορισμό της απάτης, διότι στο σχέδιο εγγράφου που λάβατε και εσείς για την καταπολέμηση αυτήν, δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης των συστημάτων πληροφορικής ιδίως του RAS, Rapid Alert System γιατί αυτό το ΡΑΣ μέχρι τώρα νομικά αφορά μόνο σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί κάποιο νομικό σύστημα και σκεφτόμαστε και το θέμα των εμπορευαμένων, των traders. Μερικοί έχουν απλώς έναν υπολογιστή, αγοράζουν ένα προϊόν και το ξαναπολούν, είτε είναι ζάχαρη είτε είναι δημητουριακά και κερδοσκοπούν βέβαια επί του προϊόντος. Είναι πραγματικά traders δηλαδή, δεν βλέπουν ποτέ το προϊόν. Και η νομική του, το νομικό του καθεστώς είναι ασαφές. Άλλα κράτη τον παίρνουν υπόψη, άλλα όχι. Και αυτό προσπαθούμε να το αποσαφηνίσουμε. Άλλο θέμα στο action plan είναι η συνεργασία, η δικαστική συνεργασία. Η Ευρωπόλ και η Ευρωζούστ, όπως ξέρετε, έχουν δικαιοδοσία εναρμόνισης των διώξεων. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο και λεπτό θέμα, γιατί πρέπει να εφαρμοστούν πάρα πολλοί νομικοί κανόνες, αλλά αφήνουμε στην Ευρωπόλ το καθήκον του συντονισμού των ερευνών έτσι ώστε όπως είπε και η κυρία Οκόνη, γέλος στο ακροατήριο, όταν υπάρχει κάποιος απατεών σε ένα κράτος μέλος να μπορεί να διωχθεί και από άλλο κράτος μέλος. Αυτό γίνεται όλο και πιο συχνά στην ενιαία αγορά. Πρέπει να μπορούν να διώκονται οι απατεώνες σε μια χώρα μέλος ακόμη και αν διέπραξαν την απάτη του σε άλλο. Και αυτό το επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπόλ. Τώρα οι κυρώσει και τα πρόστιμα. Ξέρετε ότι εδώ είναι θέμα όπου τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να δώσουν να χορηγήσουν κυριαρχία και πάντοτε αρνούνται προς την Κομισιόν εκτός αν πρόκειται για το περιβάλλον πάντοτε αρνούνται να στην Κομισιόν να τους προτείνει τα επίπεδα προστήμων ή φυλάκισης που πρέπει να επιβληθούν. Στον μελλοντικό κανονισμό εμείς λέμε ότι οι ποινές πρέπει να είναι και αποτρεπτικές αλλά τουλάχιστον να αντιπροσωπεύουν και την χρηματική αξία της απάτης ώστε όπως είπε και η κυρία Οκόνη γέλος και πάλι να υπάρχει αναλογικότητα μεταξύ της γυναίκας που κλέβει ένα μπιφτέκι και του απατεώνα που έχει αποκερδίσει πολλά. Είναι βέβαια δύσκολο το θέμα και ίσως να λυθεί αν δημιουργηθεί αυτός ο μελλοντικός Ευρωπαίος εισαγγελέα που μέχρι στιγμής πάντως είναι πολύ δύσκολο να το χειριστούμε. Θα το αναφέρει όμως ο μελλοντικός κανονισμός. Μερικοί από εσά ανέφεραν επίσης το πρόβλημα των σχεδίων ελέγχου που πρέπει να δημιουργηθούν. Σε αυτό το μελλοντικό κανονισμό για τον ελέγχους προβλέπουμε και τη δυνατότητα η Κομισιόν να επιβάλλει έλεγχο στα κράτη-μέλη γιατί σήμερα είναι μία απλή σύσταση. Τα προγράμματα ή σχέδια ελέγχου για το DNA ή το φενιλμπουταζόνιο έχουν εφαρμοστεί όταν έχουν εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη αλλά τότε υπήρχε κρίση και πήγουσα κατάσταση. Εμείς θέλουμε να έχουμε τη δυναμική δυνατότητα να οργανώνονται τέτοιοι έλεγχοι υποχρεωτικά μετά από διαβούλευση βέβαια με τα διαφορα κρατη κράτη-μέλη τακτικά ώστε να δοκιμάζονται οι διάφορες διατροφικές απάτες. Ξέρετε ότι συμβαίνουν σε πολλούς τομείς δηλαδή αντικατάσταση ενός προϊόντος από άλλο φθηνότερο, όπως αυτή η ιστορία του ολογίσιου κρέατος. Καμιά φορά το ελαιόλαδο αντικαθίσταται από, ελαιο, από κραμβέλαιο και υπάρχουν και απάτες στην ονοματολογία και σήμανση. Άλλα προϊόντα λέγονται βιολογικά ενώ δεν είναι. Και βέβαια το κέρδος είναι εδώ το κύριο κίνητρο. Ευχαριστώ τον κύριο Στάς για τις, τους επένους του για την κτηνιατρική υπηρεσία και διατροφική που είναι σημαντικό στοιχείο γιατί εκείνο θα επαληθεύει πώς εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη τα προβλεπόμενα για τις απάτες. Σήμερα έχουμε λύσει το πρόβλημα της μικροβιολογικής μόλις σαλμονέλα κλπ και τα κράτη-μέλη ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να αποφεύγουν τέτοιες μολύνσεις. Λύσαμε επίσης το θέμα της χημικής μόλυνσης με τα ανώτατα όρια για τα παρασιτοκτόνα κλπ. Και εκεί ξέρουν τα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνουν, αν και δεν το κάνουν πάντα. Αλλά για τις απάτες δεν έχουν γίνει πολλά. Και γι' αυτό ο Επίτροπος Μπόρντ θέλει να δημιουργήσει μία ομάδα απάτης σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να συντονίζονται οι έρευνες περί απατών. Σε συνεργασία και με την Όλαφ βέβαια, τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, επιχειρήσεων και άλλα καθώς και τις διάφορες υπηρεσίες όπως Ευρωπόλ και Ευρωζούστ. Γιατί αλλιώς υπάρχει κατακαιρματισμός της εργασίας μεταξύ των υγειονομικών ελεγκτών της αστυνομίας και των τελωνίων από τη μία και των εισαγγελέων ή της δικαιοσύνης από την άλλη. Πρέπει να μπορέσουμε να καταφέρουμε να συνεργαστούν όλοι αυτοί οι τομείς γιατί σήμερα στο ίδιο κράτος μέλος αλλά και σε ολόκληρη την Ένωση δυστυχώς υπάρχει πολύ κατακαιρματισμός. Τεράστιο θέμα και, και που σχετίζεται και με άλλα όπως είπε και ο κύριος Ρώση υπάρχει το θέμα της σπατάλης τροφίμων η σήμανση επίσης, όσο οι ετικέτες είναι πιο λεπτομερείς και σαφείς, τόσο λιγότερο εύκολη γίνεται η απάτη. Και ο Πίτροπος Μπόρτζ έχει αναλάβει δέσμευση να υποβάλει έκθεση τον Οκτώβριο για τη σήμανση, την προέλευση των κρεάτων. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για, που είναι υπεύθυνη για τη σήμανση των οπών κρεάτων εκτός του βοηού που έχει ήδη γίνει, των υπολείπων και πουλερικών. Αυτά θα τα κάνει συνάδελφοί μας της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και εμείς θα αναλάβουμε το θέμα της σήμανσης των κρεάτων ως συνθετικών στοιχείων ε, προετοιμασμένων πιάτων όπως λαζάνια κλπ και τον Οκτώβριο θα σας έρθουν όλα αυτά. Εδώ κύριε Πρόεδρε τι μπορούμε να σας πούμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η συγκήτρια για να κλείσουμε 30 δεύτερα. Ε, έχουμε πρόβλημα χρόνου. Ναι. Ε, δεν θα σας κάνω άλλο να υδρώνετε γιατί έφυγε ο μόνος που μου έκανε άμεση ερώτηση. Ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Θα τα ξαναπούμε, μην ανησυχείτε. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε ακόμα χρόνο για να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Καλά, η κυρία Ντελάγκη είναι πολύ πιστική. Ποιος να τολμήσει να της κάνει ερώτηση. Λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε εδώ την έκθεσή μας. Αυτή προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 27 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε κατά πάσα πιθανότητα τον Νοέμβριο. Έτσι δεν είναι. Στις 5 Νοεμβρίου, ο κύριος Σλούτερ, και στην Ολομέλεια δεν ξέρουμε ακόμα πότε. Αυτά. Τελειώνει η συζήτηση για αυτό το θέμα και σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Και τώρα, ερχόμαστε στο σημείο 19. Επενδύσεις στην υγεία. Τώρα όμως θα δώσω το λόγο στην κυρία Τεστόρη, τη Γενική Διευθύντρια, για να μας κάνει αυτή την εισαγωγή της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης ε, που δεχτήκατε να εντάξετε τώρα αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Γιατί το ζητήσαμε. Διότι θέλουμε να επιμείνουμε στη σημασία που έχει το γεγονός ότι ε, η υγεία η υγεία δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του κράτους, αλλά και ως επενδυτική ευκαιρία που μπορεί να δώσει μερίσματα και να πληρώσει στην κοινωνία. Ε, είναι τμήμα τώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θα ξέρετε, η υγεία. Πριν από λίγες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις συστάσεις αναχώρα και είναι 11 πλέον τα κράτη-μέλη που ε, έχουν στις συστάσεις τους ζητήματα που αφορούν την υγεία γενικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να κοιτάξουν την μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας τους έτσι ώστε να είναι ε, αποτελεσματικό το κόστος, δηλαδή οικονομικό. Τι, τι εννοούμε, γιατί το λέμε αυτό. Θέλουμε να έχουμε συστήματα υγείας που να χρησιμοποιούν τους δημοσίους πόρους με τρόπο αποτελεσματικό μεν, αλλά και ταυτόχρονα να παρέχουν πρόσβαση σε ποιότητα υψηλή ε, υπηρεσιών υγείας. Αυτή τη στιγμή που η διαχείριση των συστημάτων υγείας είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των κρατών ε, μελών, αυτοί οι καιροί έχουν παρέλθει. Διότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη τα εθνικά συστήματα υγείας έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομία τους, στο ε, προϋπολογισμό τους και στα δημόσια οικονομικά, άρα και στην οικονομία των υπολείπων κρατών μελών. Ε, θεωρούμε ότι η υγεία είναι μια αξία αυτή καθ' αυτή, αλλά είναι και κομβικό στοιχείο για μια οικονομική επιτυχία. Οι δαπάνες υγείας, αν είναι αποτελεσματικές και εύστοχες, Ε, συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Είναι θετικές δαπάνες άρα. Λοιπόν, εμείς στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ε, έχουμε εκπονήσει αυτό το χαρτί που ονομάζεται επένδυση στην υγεία και καλώ όλους τους ευρωβουλευτές να το διαβάσουν γιατί για αλλαγή είναι πραγματικά, είναι πολύ καλό το έγγραφο, διαβάστε το, αξίζει τον κόπο, να το πείτε στους συναδέλφους σας πρόεδρε κοιτάζει την επένδυση στην υγεία από ένα τριπλό πρίσμα. Πρώτον, όταν επενδύεις στην υγεία, τι επιτεχάνεις. Αηφορία και βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, οπότε και καλύτερη εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών των κρατών μελών. Είναι σαφές ότι υπάρχουν προκλήσεις ε, στα συστήματα υγείας μας σήμερα και μεγάλες. Ο πληθυσμός γυράσκει είναι μεγάλο και το κόστος και το βάρος από τις χρόνιες ασθένειες, άρα όλο και περισσότερο υπάρχει ζήτηση για υπηρεσίες υγείας για περίθαλψη, όλο και περισσότερο αναζητούνται νέες τεχνολογίες και νοτόμες, αλλά έχουμε όλο και λιγότερα χρήματα ή χρειάζεται εξυγίαση και ο προϋπολογισμός της υγείας διότι το ταμείο είναι μείον. Ε, χρειάζεται λοιπόν να αυξηθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων και η αποδοτικότητα και όταν προτείνουμε οικονομίες στον προϋπολογισμό της υγείας δεν εννοούμε ξερές δαπάνες, στεγνές, αλλά ε, δαπάνες που κοιτούν και το μέσο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει εδώ τα κράτη-μέλη. Πρώτον, η οδηγία για τη διασυνοριακή περίθαλψη εφαρμόζεται και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και γνώση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη τα συστήματα υγείας, τι δικαιώματα έχουν οι ασθενείς στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία, τι γίνεται με τις κλινικές ε, δοκιμές και πληρονομοσύνες και γενικά πώς εφαρμόζεται αυτή η οδηγία. Επίσης βοηθούμε τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συγκεντρώνουμε τους πόρους μας για την τεχνολογική υγεία, για την ηλεκτρονική υγεία, το e-health, έτσι ώστε να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη και να προοδεύουν στην κατεύθυνση αυτή. Ε, επίσης, έχουμε συστήσει ένα πάνελ ε, εμπειρογνωμόνων για την πραγματογνωμοσύνη από τα κράτη-μέλη και επίσης συνεργαζόμαστε με τον συνάδελφο που είναι αρμόδιος για τα διαρθωτικά ταμεία να βοηθήσει τα κράτη-μέλη ε, έτσι ώστε να εντάξουν στα εθνικά τους προγράμματα την επένδυση στην υγεία αλλά με τρόπο σωστό και αποτελεσματικό. Δεύτερη προτεραιότητα του εγγράφου μας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αν επενδύουμε στην υγεία ε, έχουμε καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό. Να σας δώσω μια ιδέα. Με ποιο τρόπο η υγεία, ε, μάλλον 3 με 6% ε, του χρόνου εργασίας χάνεται γιατί λείπουν οι εργαζόμενοι από τη δουλειά τους για λόγους υγείας, που σημαίνει αυτό 2% του ΑΕΠ. Δηλαδή, ε, αν βελτιωθεί ε, η υγεία των εργαζομένων, θα εργάζονται πιο αποτελεσματικά και δεν θα απουσιάζουν από τη δουλειά τους για λόγους υγείας. Άρα είναι κέρδος αυτό. Επίσης, όταν μιλούμε για επένδυση στην υγεία του ανθρωπίνου κεφαλαίου, αυτό προάγει και τη δημόσια υγεία, δεν θεραπεύει μόνο. Τα κράτη-μέλη επικεντρώνονται πάρα πολύ στη θεραπεία και πολύ λίγο στην πρόληψη και στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Τρίτο σημαντικός πυλώνας αυτού του εγγράφου μας, στην επένδυση στην υγεία, είναι οι ανισότητες στην υγεία. Επενδύοντας στην υγεία μειώνουμε τις ανισότητες που επικρατούν και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγον αυτό για ε, την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση αποκλεισμών. Ε, είναι μαζική σπατάλη ανθρωπίνου δυναμικού οι ανισότητες ε, στην υγεία άρα και οικονομικού ε, δυναμικού. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι να διατηρηθεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής κοινωνίας που είναι καθολική προσέγγιση σε υψηλής ποιότητας και ασφαλής υπηρεσίες υγείας για όλο τον πληθυσμό. Συμπέρασμα. η προαγωγή της υγείας, ε, τα ε, αποδοτικά ε, συστήματα υγείας είναι σημαντικό να τα βλέπουμε και από την οικονομική σκοπιά. Δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε την αξία που αρμόζει στην υγεία, αλλά θέλουμε να αποδείξουμε ότι η υγεία είναι και παράγον της οικονομίας και μάλιστα κινητήρια δύναμη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τεστόρη. Ο κύριος Πέτερλε έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Πρέπει να σας πω ότι ότι λέγω δεν με βρίσκουν σύμφωνο οποιασδήποτε πρωτοβουλίες της Κομισιόν αλλά δύο πράγματα με ικανοποιούν η συνεργασία για την καταπολέμηση του καρκίνου μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου άρχισε η Κομισιόν αυτό, άνοιξε το νέο αυτό μέτωπο και το δεύτερο σημαντικό είναι η πρωτοβουλία την οποία συζητάμε σήμερα που και αυτή με ικανοποιεί αυτή με ικανοποιεί για τον φιλοσοφικό λόγο στον οποίο οφείλεται. Δηλαδή θέλω να δω σε τι αξίες βασίζει την αντίδραση της η Κομισιόν. Την υγεία δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε σαν ένα οποιονδήποτε οικονομικό τομέα. Είναι και κοινωνικό θέμα όχι μόνο για τον διαβήτη και τον καρκίνο, αλλά και γενικότερα. Και η εντύπωσή μου είναι ότι η κρίση αυτή του υγειονομικού μας συστήματος θα κρατήσει παραπάνω από τη χρηματοπιστωτική. Ελπίζουμε αυτή η τελευταία να, αρχί, να έχει αρχίσει να τελειώνει. Αλλά η φιλοσοφία αυτή της αλληλεξάρτησης που αποδείχτηκε και για το χρηματοπιστωτικό τομέα ισχύει και στα υγειονομικά. Εγώ είμαι υπέρμαχος βέβαια της επικουρικότητας, νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε τις συνθήκες, αλλά υπάρχουν και θέμα που δεν μπορούν να θέματα που δεν μπορούν να λυθούν μόνο με την ε, δήλωση ότι τα υγειονομικά είναι θέματα των χωρών μέλων. Κανένα καμία χώρα μέλος δεν μπορεί από μόνη της να τα λύσει όλα αυτά αλλά μόνο σε υψηλότερο επίπεδο και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κομισιόν το τονίζει. Βλέποντα τα μέτρα αυστηρότητας που επιβάλλονται και στον τομέα της υγείας, τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις τους την χάνουν και δικαίω επικρίσεων γιατί τα θεωρούν σαν απλή εξοικονόμηση και όχι και αγνοούν το ότι μπορεί να χειροτερεύουν έτσι την υγεία του ανθρώπινου κεφάλαιου. Εδώ υπάρχουν πολλές νέες δυνατότητες για να κάνουμε κάτι. Αν αναγνωρίσουμε δηλαδή ότι θα καταφέρουμε πολλά περισσότερα με συνεργασία. Αν εκμεταλλευτούμε καλύτερα την υπάρχουσα γνώση και πληροφόρηση, τότε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και να μειώσουμε και τις ανισότητες. Είναι λοιπόν νομίζω πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή. Δεν σας κάνω ένα πολιτικό κομπλιμέντο. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι καθεαυτού σωστό και νομίζω ότι καλό είναι να τονίσουμε περισσότερο την πρόληψη. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να υπάρχουν υπουργεία πρόληψης στα κράτη-μέλη. Γιατί αν επενδύσουμε σε αυτήν, τότε θα αλλάξουν τα πράγματα δραματικά. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη. Είναι πολύ καλή επένδυση. Ευχαριστώ πολύ. και Σλούτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που μόλις είπε και ο συνάδελφος επενδύσεις στην υγεία. Ένα θέμα πολύ σημαντικό, το ίδιο και η παιδεία, οι καλές ε, καθημερινές συνήθειες, και το βιωτικό επίπεδο. Εάν θέλουμε μια υγιή κοινωνία στην Ευρώπη, εάν εξασφαλιστούν αυτά, τότε και μόνο τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε και για μεταρρύθμιση των υγειονομικών μας συστημάτων, των συστημάτων πρόνοιας, το πώς ε, θα βελτιωθούν ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ήθελα να σταθώ και στο σημείο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Αυτό είναι κάτι που συχνά το επαναλαμβάνουμε στην Επιτροπή μας. Η πρόσβαση στις καλές υγειονομικές υπηρεσίες πολλές φορές εξαρτάται απλώς και μόνο από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Βεβαίως, σημαντικό είναι και να επαληθεύσουμε και να παρακολουθούμε πώς ε, εξελίσσεται αυτή η διαδικασία ώστε να εξαλείψουμε τις ανισότητες στα υγειονομικά συστήματα ιδίω σε αυτόν τον τομέα που είναι άκρος ιατρικού χαρακτήρα για υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες για χρόνιες παθήσεις και για πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Θα έλεγα ότι ίσως πρέπει να αντιστραφούν και οι προτεραιότητες. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως μόλις είπε ο συνάδελφος, είναι η πρόληψη, η πρόληψη και ξανά άλλη μια φορά πρόληψη. Τι θα κάνουμε δηλαδή για τις επόμενες γενναίες. Το μέλλον πρέπει να φροντίσουμε, ώστε οι μελλοντικές γενναίες να μην χρειαστεί να χρησιμοποιούν το σύστημα υγείας στο βαθμό που εμείς το χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε κύριε Σλίτερ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλό να συζητήσουμε με τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και άλλους που θέλουν να καταστρέψουν με χημικές ουσίες και άλλα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, να καταστρέψουν το σύστημα υγείας μας. Ελπίζω στην ανακοίνωσή σα να εξηγήσετε και στι άλλε γενικέ διευθύνσει πόσο σημαντικά είναι αυτά και θα προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και εμεί το ίδιο ε, το Κοινοβούλιο και τι ενδιαφερόμενε επιτροπέ για την οδηγία για το κάπνισμα λόγω χάρη και τα προϊόντα καπνού. Βλέπουμε πώ το αντιμετωπίζουμε εμεί ενώ συζητιέται στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντο, μάλλον σε άλλη επιτροπή συζητιέται πώ να ενισχυθεί η οδηγία αυτή. Έχουμε πολύ διαφορετικέ απόψει και προσεγγίσει κάποιε φορέ. Νομίζω το ίδιο όπω και με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και την Τρόικα. Ζητούν από την Ελλάδα να μειώσουν τι δαπάνε τη υγεία. Ανησυχώ για τέτοιου είδου συστάσει. Ε, πρέπει να υπάρχει μια σαφή πολιτική. Να, τι είπατε κι εσεί τώρα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με, στο επίπεδο όλων των θεσμικών οργάνων. Ή για του μηχανισμού κοινοτομία και την εξοικονόμηση κονδυλίων για την υγεία. Τα ειδικά ταμεία. Τα ταμεία αυτά Τα price funds λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, μόνο σε ειδικέ περιπτώσει, όπω έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με μικρά κονδύλια, περιορισμένου πόρου από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό μπορούμε να κάνουμε τεράστια επιτέγματα, μπορούμε να έχουμε τεράστια επιτέγματα, όπω την έρευνα. Και η γενική μας ε, θεώρηση της κοινωνίας, διαρκής ε, πίεση για ανάπτυξη, για περισσότερη δουλειά στους εργαζόμενου, αυτό επηρεάζει και την υγεία των ανθρώπων. Η προσωπική μου σταυροφορία εδώ είναι να μειώσουμε το χρόνο εργασία αυξάνοντα την αποτελεσματικότητα. Όχι να αυξάνουμε την παραγωγή και να δημιουργούμε μόνο έτσι, με ένταση ε, νέε θέσει εργασία. Και του ανθρώπου θα εξαντλήσουμε έτσι και του πόρου, προσπαθώντα να δημιουργήσουμε θέσει εργασία. Είναι άλλο το θέμα βέβαια, αλλά νομίζω ότι καλό ήταν να ακουστεί και εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλει η Γενική Διευθύντρια να ξαμιλήσει, να απαντήσει σε ερωτήσεις ε, που έγιναν, παρακαλώ κυρία Τεστόρη. Ναι, λίγα πράγματα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πρώτον, χαίρομαι και ε, εκτιμώ αυτό που είπε ο κύριος Πέτρελε για την επικουρικότητα. Είναι σαφές ότι σεβόμαστε ε, την επικουρικότητα, αλλά συμφωνώ με τον άλλο εις ότι δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα των καλύτερων συστημάτων υγεία στα κράτη-μέλη αν δεν συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και τους πόρους μας. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Για την κυρία Χίμπνερ, συμφωνώ. Η προαγωγή υγείας, πρόληψη ε, της υγείας είναι κάτι το οποίο δεν απασχολεί αρκετά τα κράτη-μέλη. Εκεί δίνουμε τη μάχη μας. Και σε σχέση με τον κύριο Σλούτερ, είναι κοινό ο αγώνας, αλλά ε, ε, το δικό μας έγγραφο επένδυση στην υγεία είναι το σώματος των επιτρόπων. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι η υγεία δεν συνιστά δαπάνη αλλά επένδυση. Και το θέμα της μεγαλύτερης παραγωγικότητας και ε, της καλύτερης απόδοσης του εργατικού δυναμικού ε, προσπαθώ να καταπολεμήσω την απουσία από την εργασία λόγω ασθενείας. Δηλαδή, αν έχουν καλύτερη υγεία εργαζόμενοι, θα κάνουν κανονικά τη δουλειά τους με καλύτερο τρόπο και δεν θα λείπουν. Δεν είναι αύξηση της παραγωγικότητας, είναι ε, αποφυγή ε, απουσίας από την εργασία λόγω ασθενείας. Ευχαριστώ που μας ακούσατε και μας δεχτήκατε για αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τεστόρη. Λοιπόν, θα διαβάσουν οι συνάδελφοι αυτό το έγγραφο. Θα επιθυμούσαν είναι και περισσότεροι παρόντες, γιατί το έγγραφο το αξίζει. Ε, θα συνεχίσουμε όμως την προσπάθεια, θα το παρακολουθήσουμε, δεν θα το παραμελήσουμε. Είναι σημαντικό θέμα υγεία και μόνο μια υγεία την έχουμε και μόνη. Ε, μάλιστα. Και το καταλαβαίνουμε όταν τη χάνουμε αυτό κυρίως. Ε, επόμενη συνεδρίαση για εξαίρεση στο Στρασβούργο παρακαλώ 4 Ιουλίου 9 με 12 το μεσημέρι απευθύνομαι στους συναδέλφους που παρευρίσκονται να πάρετε και να έχετε μαζί σας κάρτες ψηφοφορίας και 10 και 11 Ιουλίου μαραθώνιος θα είναι όπως δεν τον έχετε ξαναζήσει ποτέ στη ζωή σας θα ψηφίσουμε για τα καπνά και ενδεχομένω για τα ιατροτεχνικά προϊόντα και άλλα τεινά ενδιαφέροντα. Να βαρεθείτε, αποκλείεται. Χθε ήταν μόνο μία πρώτη γεύση για το τι σας περιμένει. Λοιπόν, 10 και 11 Ιουλίου, μην κανονίστε τίποτα άλλο, κρατήστε οπωσδήποτε ελεύθερη τη μέρα γιατί ψηφίζουμε αγρίως. Και στι 4 Ιουλίου στο Στασβούργο, λήξη συνεδρίαση. καλή σας ε, επιστροφή και να είστε καλά. Χαίρετε.